Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήλθατε στη συνεδρίασή μας. Να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις για την ημερήσια διάταξη. Ε, καταρχήν, να ζητήσω αν έχετε αντιρρήσεις, εάν όχι θεωρείτε δεδομένη δεκτή η ημερήσια διάταξη. Και επίσης, έχετε διάφορα στοιχεία στο έγκυρο έντυπο Cont News σε σχέση με τις γλώσσες εργασίας, τις γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούνται για διερμηνία και όπως ξέρετε η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο μέσω web streaming. Και έχουμε τώρα στο σημείο 3 της σημερισίας διάταξης. Έγκριση των πρακτικών μας της 18 και 19 Φεβρουαρίου και επίσης 21ης Φεβρουαρίου Έχετε εδώ αιτήσει για τροποποιήσει, ή αντιρίσει, ή αντιρρήσει, εάν όχι. Θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί λοιπόν τα πρακτικά και περνάμε κατευθείαν στο σημείο 4, την κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Πρόκειται για την ε, εξέταση ενός σημαντικού θέματος που είναι η παρουσίαση της μελέτης για την υποστήριξη στον προϋπολογισμό. Το ερώτημα είναι κατά πόσο και με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο ανάπτυξης. Χαίρομαι για την παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης, της κυρία Ζολή, η οποία και αυτή μπορεί να μας παρουσιάσει την ε, το περιεχόμενο αυτό της έκθεσης. Για μας ως Επιτροπή Ελέκτου Προπολογισμού μας ενδιαφέρει όταν εμπλέκονται χρήματα φορολογουμένων πώς στην πράξη αποδίδουν καρπούς. Αυτό το εργαλείο λοιπόν, η υποστήριξη προς τον προϋπολογισμό είχε σταθεί στο παρελθόν αμφιλεγόμενη, αλλά είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι συνδέεται αυτή η χρήση αυτού του εργαλείου με τη διατήρηση των καταλήλων αρχών στις χώρες ανάπτυξης, ότι συνδέεται με ευκυβερνησία και διαφάνεια. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσο αυτά τα μέσα τελικά έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα ή όχι. Αυτό είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, διότι σε πολλές ε, χώρες έχουν γίνει μέσω αυτής της έρευνας μελέτες για τον αντίκτυπο και το αποτέλεσμα που έχουν αυτές οι μορφές ε, υποστήριξης, του προπολογισμού. Αυτά ήθελα να πω εγώ και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ζολή. Καλώς ήλθατε φυσικά και χαίρομαι που θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση και ελπίζω δεν είναι τελευταία ευκαιρία αυτού του είδους. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και των άλλων επιμέρους επιτροπών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ σήμερα να συμπροεδρεύσω σε αυτή τη συνεδρίαση που θα εξετάσουμε μία έκθεση που ετοίμασε ένα από τα κράτη-μέλη, οι κάτω χώρε για την δημοσιονομική στήριξη. Όπως θα γνωρίζετε, η δημοσιονομική στήριξη είναι μια πολύ συνήθις μορφή αναπτυξιακής βοήθειας. Αφορά περίπου το 1 τρίτο των κονδυλίων του μέσου που διαθέτουμε, του ECI, και το 75% παγκοσμίω τη βοήθεια που παρέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε κατά πόσον το εργαλείο αυτό είναι αποτελεσματικό, πλήρω αποτελεσματικό και αυτό είναι κάτι που συζητιέται ευρέω σε πολλέ χώρε. Χωρί λοιπόν να καθυστερήσουμε περαιτέρω, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Αντουάν Ντεκέμπ. Κύριε Ντεκέμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ονομάζομαι Άντωνη Ντεκέμπ και εργάζομαι για το Τμήμα Αξιολόγησης Πολιτικών και Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της ε, Ολλανδικής Κυβέρνησης. Πέρυσι κάναμε μια αναθεώρηση της πολιτικής για τη δημοσιονομική στήριξη και αναλύσαμε τις Ολλανδικές πολιτικές για τη δημοσιονομική αυτή στήριξη, αλλά δεν θα σας δώσω περιττές λεπτομέρειες για αυτό το τμήμα της μελέτης σήμερα το απόγευμα. Απλώς θα προσπαθήσω να δω τι γνωρίζουμε πραγματικά, να παρουσιάσω τι γνωρίζουμε για την ε, δημοσιονομική στήριξη, για την αποτελεσματικότητά της, το πώς λειτουργεί. Όπως υπόθηκε, είναι ένα αμφιλεγόμενο μέσο και ιδίως στις κάτω χώρες. Και σήμερα το πρόγραμμα, το απόγευμα, Θα ήθελα να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Να δούμε πώς θα μπορούσε ή μπορεί να λειτουργεί η δημοσιονομική στήριξη. Για αυτό το σκοπό καλό θα ήταν να δούμε κάποια ιστορικά δεδομένα. Εάν δείτε τι έγινε σε προηγούμενες δεκαετίες, σε χώρες πολύ χαμηλού εισοδήματος, εκεί δεν υπήρξε σοβαρή βελτίωση στο εισόδημά τους, όπως βλέπετε με τη γαλάζια γραμμή στο διάγραμμα. Στο κάτω μέρος της γραφικής παράστασης. Αρχικά η Αφρική τα πήγαινε κάπως καλύτερα, αλλά από, τα... από τη δεκαετία του 80 και μετά το 90 όταν είχαμε την προηγούμενη οικονομική κρίση, τα επίπεδα του εισοδήματος στις περισσότερες αφρικανικές χώρες μειώθηκαν. Εάν δείτε την πράσινη γραμμή, τη Ζάμπια δηλαδή, εδώ βλέπετε ένα ακραίο παράδειγμα. αποτέλεσμα κακής οικονομικής διαχείρισης του τι, πώς χειρίστηκαν τα ορυχεία χαλκού και των τιμών βεβαίως στη διεθνή αγορά. Η Ζάμπια δεν τα πήγε καλά. Το εισόδημα έπεσε. Ε, υπήρξε τεράστια σώρευση χρέους και τα χαμηλά επίπεδα εισοδήματος σε συνδυασμό με τους υψηλούς τόκους ανάγκασαν την κυβέρνηση να μειώσει τις δαπάνες ε, των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχονταν. Όπως θα δείτε και στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε ένα μικρό κοινοτικό σχολείο στο βορρά της χώρας. Και εδώ αυτό που ήθελα σε εσά να πω σήμερα το απόγευμα είναι ότι εγώ αυτό το κορίτσι το γνώρισα. Ήταν εθελόντρια σε ένα σχολείο, δασκάλα που δίδασκε σε δύο τάξεις. Σε ένα σχολείο 169 μαθητών, μόνη τη. Εδώ λοιπόν το θέμα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα τέτοιο κορίτσι που δεν είναι το επαγγελμά του ακριβώς να είναι δασκάλα, μόνο με συγκεκριμένα προγράμματα. Και τι γίνεται με το διπλανό σχολείο, το γειτονικό. Εδώ υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα. Έτσι, ως δωρητές, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πολλά παράλληλα προγράμματα. Όμω το ερώτημα είναι θα ήταν κάτι τέτοιο αποτελεσματικό. Εδώ έρχεται να προσφέρει κάτι η δημοσιονομική στήριξη. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα το απόγευμα να σα παρουσιάσω την πολιτική θεωρία για την δημοσιονομική στήριξη, τη μεθοδολογία που ακολουθούμε. <clears throat> Μην ανησυχείτε, θα είμαι πολύ σύντομο για αυτό το σημείο. Τα άμεσα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο στην διακυβέρνηση ιδίω, τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη και κάποια συμπεράσματα τα οποία θα ήθελα να, στα οποία θα ήθελα να καταλήξω. Όπως ξέρετε λοιπόν για την δημοσιονομική στήριξη, είναι μια απευθείας ροή ε, κονδυλίων στην κυβέρνηση της δικαιούχου χώρας, η οποία συνοδεύεται από διάλογο για πολιτικές μεταξύ κυβέρνησης και δωρητών, και συνήθως είναι μια πολυμερή συζήτηση με πολλού ε, δωρητέ. Στη λόγου χάρη, Συμμετείχαν 19 δωρητέ. Τώρα ε, βέβαια 100 χώρε αποσύρθηκαν πέρσι, οπότε έχουν μείνει 18. Και στην Τανζανία μιλάμε για 14 δωρητέ αυτή τη στιγμή. Πολλοί λοιπόν από του δωρητέ, ε, είναι πολλοί συνήθω οι δωρητέ που παίρνουν μέρο ταυτόχρονα στο ίδιο πρόγραμμα δημοσιονομική στήριξη. Τώρα, γιατί δημιουργείται ένα τέτοιο εργαλείο, ένα τέτοιο μέσο, Γιατί δεν υπάρχει αρκετή αποτελεσματικότητα ή βιωσιμότητα των ε, προγραμμάτων. Επίσης υπάρχει απογοήτευση με την εξάντη αιρεσιμότητα. Τα προγράμματα δηλαδή που είχαν ε, καταρτιστεί στη δεκαετία του 80 και του 90. Εάν δείτε τι γινόταν τότε, οι κυβερνήσεις δικαιούχοι έπαιρναν χρήματα αφού υπόσχονταν ότι θα βελτιώσουν τις πολιτικές τους, ιδίως τις οικονομικές. Όμως η εμπειρία και η αξιολόγηση εκ των υστέρων έδειξε ότι αυτή η ρασιμότητα τελικά δεν ήταν αποτελεσματική. Ανταυτού λοιπόν, αντί να προσφέρονται χρήματα βάσει υποσχέσεων, ουσιαστικά, αντιστρέψαμε τα πράγματα. Οι κυβερνήσεις έπαιρναν χρήματα πλέον, έπαιρναν κονδύλια, όταν ήδη εφάρμοζαν κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές, στρατηγικές για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και η Παγκόσμια Τράπεζα είχε εκπονήσει εκθέσεις που έδειχναν ότι χώρες με καλές πολιτικές με καλές μακροοικονομικές πολιτικές τα πήγαιναν πολύ καλύτερα ως προς την οικονομική τους αύξηση από ότι χώρες με πολιτικές που ήταν χάλια. Τέλος, έπρεπε να αποδεχτούμε ότι, ότι αν θέλαμε να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη, ήταν επιτακτική ανάγκη να συνεργαστούμε στενά με κυβερνήσεις και με τις δομές των κυβερνήσεων. Λόγου χάρη για τη δημοσίευση δικτών, για την υγεία. Υπήρχε η αίσθηση ότι η δημοσιονομική στήριξη θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια πιο εναρμονισμένη, πιο προβλέψιμη, να ε, βελτιώσει τη μείωση του κόστους των συναλλογών, να οδηγήσει σε ανάληψη ευθύνης από τους δικαιούχους και να είναι πιο αποτελεσματική η προσφορά βοήθεια. με πιο βιώσιμα αποτελέσματα. Αυτό στα τέλη τη δεκαετίας του 90 και τι αρχέ της νέας χιλιετίας. Έτσι, η δημοσιονομική στήριξη αυξήθηκε από 1,9 δις το 2002 σε 5,3 δις το 2009. Μιλάμε πάντα για αμερικανικά δολάρια. Εάν δείτε τα δικά μας δεδομένα για τις κάτω χώρες, εμείς προσφέραμε σε μια περίοδο δεκαετίας 1,75 δις ε, δημοσιονομικής στήριξης, γενικής δημοσιονομικής στήριξης, περίπου, όχι βέβαια ένα τρίτο του δικού μας προπολογισμού, αλλά 3,4% για την αναπτυξιακή συνεργασία. Δεν ήταν και πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και όμως οι κάτω χώρε ήταν ένας από του μεγαλύτερου δωρητέ για την δημοσιονομική στήριξη, μέσα με χώρε όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Νορβηγία και βεβαίως η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις δικαιούχες χώρες ήταν λιγότερο από 3% του ΑΕΠ τους ε, η προσφορά αυτή. Και σε πολλές από αυτές λιγότερα από 6 ευρώ ανακάτοικο ετησίως. Εάν θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής στήριξης και να τα αξιολογήσουμε, πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Εάν δούμε τις αρχικές πολιτικές θεωρίες, όπως, τις έχω, και εγώ, όπως έχω προσπαθήσει να τις ε, απεικονίσω εδώ, η βασική ιδέα ήταν ότι θα έπρεπε να έχουν σταθερέ οικονομικέ πολιτικέ κυβερνήσει να λειτουργούν ώστε να μπορούν να επιλεγούν και να του αποδοθεί δημοσιονομική στήριξη. Έπειτα πιστεύαμε ότι η δημοσιονομική στήριξη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάληψη της ευθύνης και αποτελεσματική καταπολέμηση της φτώχειας και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, πιο σταθερά αποτελέσματα. Αυτή ήταν η αρχική θεωρία. Όμως, πολύ γρήγορα, οι δωρητές άρχισαν να μεταβάλουν τη θεωρία αυτή. Πρώτα απ' όλα, πολλές χώρες δεν είχαν τέτοιες εύρωστες οικονομικές πολιτικές, σταθερές μακροοικονομικές πολιτικές. Οπότε αλλάξαμε λίγο τα πράγματα. Είπαμε ότι θα μπορούσε η δημοσιογραφική στήριξη να γίνει κίνητρο για να βελτιωθούν οι υπάρχουσες πολιτικές. Και πάλι ε, το στοιχείο της παλιάς ερεσιμότητας άρχισε να ξαναισχύει. Δηλαδή ένας μαζικός μηχανισμός χρηματοδότησης έγινε η δημοσιονομική στήριξη που λειτουργεί ως κίνητρο για την βελτίωση μακροοικονομικών πολιτικών. Αλλά δεν σταματάει εδώ η ανάπτυξη αυτής της θεωρίας. Ακολουθεί πέραν της αρχικής σύλληψης ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν σταθερές οικονομικές πολιτικές που ήδη να λειτουργούν, πέραν της ιδέας αυτής οι δωρητές άρχισαν να απαιτούν και καλή διακυβέρνηση, ευκυβερνησία ως μια πρώτη προϋπόθεση για να προσφερθεί δημοσιονομική στήριξη. Ο λόγος για αυτήν την αξίωση και ως κριτήριο επιλογής ήταν ε, μια προϋπόθεση, έτσι θεωρήθηκε, για την πραγματική οικονομική ανάπτυξη και την πραγματική καταπολέμηση της στόχιας. Όπως όμως τα γνωρίζετε σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, η διακυβέρνηση. Το τι κάνουν οι κυβερνήσεις και το εάν το κάνουν αποτελεσματικά δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτιμηθεί με βάση τις δικές μας, ε, τα δικά μας κριτήρια. Οπότε και πάλι μπήκε το στοιχείο των κινήτρων. Η δημοσιονομική στήριξη προσφερόταν ως κίνητρο για τη βελτίωση της καλής διακυβέρνησης, για την ενίσχυσή της. Ο διάλογος περί πολιτικών και επιλογών, ο πολιτικός διάλογος ήταν κάτι που θα έπρεπε να πηγαίνει μαζί. Ήταν λοιπόν ένα στοιχείο ερεσιμότητας, ε, ένα κριτήριο επιλογής. Η δημοσιονομική στήριξη έγινε κίνητρο για τη βελτίωση της κυβέρνησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και οι από το παρελθόν. Μια διαφάνεια γρήγορη για την μεθοδολογία μας. Είδαμε προηγούμενες αξιολογήσεις, κάποιες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημαντικές αξιολογήσεις όπως την Τινησία, είδαμε τα στοιχεία τα, τις, τα πανεπιστημιακά που υπάρχουν, τα ακαδημαϊκά στοιχεία. Ε, κάναμε κάποιες οικονομετρικές αναλύσεις για τον αντίκτυπο της δημοσιονομικής στήριξης και μετά συγκρίναμε χώρες μεταξύ τους, έξι συγκεκριμένα, την Κάνα, το Μαλί, την Ικαράγουα, την Τανζανία, το Βιετνάμ και τη Ζάμπια. Έτσι επιλέξαμε τις έξι χώρες από αυτή τη γραφική παράσταση. Με την οριζόντια πρόσβαση που μπορεί να έχουν. Βλέπετε τη δημοσιονομική στήριξη ως ποσοστό της, ε, των ε, κυβερνητικών δαπανών. Και βλέπετε στα δεξιά Τανζανία, Ρουάντα, Μοζαμβίκη, χώρες που έχουν λάβει μεγάλη δημοσιονομική στήριξη, ενώ από την άλλη, στα αριστερά, χώρες όπως τη Βολιβία, την Ικαράγουα, το Βιετνάμ, τη Σενεγάλη, που δεν έχουν λάβει και τόσο πολύ στήριξη. Ενώ στον κάθετο άξονα, στη μεσαία λωρίδα, βλέπετε το μέσο όρο τα, τη βαθμολόγηση Kaufman της Παγκόσμιας Τράπεζας για την καλή διακυβέρνηση με χώρες όπως ε, την Ουγκάντα, τη Ζάμπια, την Νικαράγουα, την Βολιβία και έτσι επιλέξαμε τις έξι χώρες από την πλευρά της Ολλανδικής κυβέρνησης. Εάν δούμε τα άμεσα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο στη διακυβέρνηση της δημοσιονομικής στήριξης, Πρώτον, βλέπουμε ότι η δημοσιονομική στήριξη επέτρεψε να βελτιωθεί η εναρμόνιση, να ενισχυθεί η εναρμόνιση. Βέβαια, από την άλλη, οι δωρητέ ακολουθούσαν τι δικέ του πολιτικέ προτεραιότητε. Θα δείτε ότι στο πλαίσιο των αποτιμήσεων επιδόσεων ήταν πολλοί οι δωρητέ, πολλοί ειδικοί ανατομέα και ο καθένα ε, έβαζε ω προτεραιότητα τα δικά του συμφέροντα ή προτεραιότητε. Η προβλεψιμότητα της βοήθειας βελτιώθηκε βαθμιδών, αλλά οι περισσότεροι δωρητές συνήθως εκταμείευαν προς το τέλος της χρονιάς. Αυτό υπήρχε, παρέμενε ένα πρόβλημα για τις δικαιούχους χώρες. Επίσης ενισχύθηκαν τα τοπικά συστήματα, ιδίω με τη χρήση των ε, κυβερνητικών δομών και υπηρεσιών, αλλά ένα από τα βασικά αποτελέσματα της δημοσιονομικής στήριξης είναι, υπάρχει εδώ σχέση αιτίου αιτιατού, ε, είναι ότι υπήρξε αύξηση των πόρων για συγκεκριμένου ε, τομεί, ιδίω του κοινωνικού. Αλλά ο αντίκτυπο ήταν περιορισμένο στην διακυβέρνηση. Για την ε, δημόσια δημοσιονομική, για την ε, δημοσιονομική διαχείριση, για, την, για άλλους θεσμούς, όπως η θέση του Γενικού Ελεγκτή. Όμως τα αποτελέσματα αυτά είναι μέτρια. Μίλησα για την καλή διακυβέρνηση ως προϋπόθεση για την επιλογή. χώρες σαν τη δική μας, όπως όλοι, κάτω δηλαδή, δημοσιονομική στήριξη προσφέρουν μόνο σε χώρες που ήδη έχουν πολύ σταθερές μακροοικονομικές πολιτικές. Εάν δούμε τις διαφορετικές χώρες και τις συγκρίνουμε, στα αριστερά βλέπετε χώρες που δεν έλαβαν μεγάλα ποσά δημοσιονομικής στήριξης, ενώ στα αριστερά το αντίθετο η διαφορά μεταξύ τους τελικά δεν είναι μεγάλη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι δωρητές ε, την καλή διακυβέρνηση τη χρησιμοποίησαν ουσιαστικά ως προϋπόθεση. Μάλιστα. Χρησιμοποίησαν τη δημοσιονομική στήριξη ως κίνητρο για τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω του διαλόγου περί πολιτικών, του πολιτικού Ποιος ήταν ο αντίκτυπος τώρα αυτών των ε, πολιτικών. Βλέπετε την, ε, ως ποσοστό του ΑΕΠ την δημοσιονομική στήριξη και βλέπετε ότι δεν είναι άμεσος ο συσχετισμός. Χώρες που έλαβαν μεγάλη δημοσιονομική στήριξη δεν τα πήγαν πολύ καλύτερα τελικά από αυτές που δεν πήραν και από τις επιδόσεις τους στην ε, διακυβέρνηση, στην ευκυβερνησία. Υπάρχουν βέβαια τρεις περιπτώσεις ε, που είναι εξαίρεση εκτός κατηγορίας. Η Ρουάντα, η Σχεραλεώνα και το Μπουρούντι. Ξεκίνησαν με πολύ χαμηλά ποσοστά ευκυβερνησίας ε, στις αρχές της χιλιετίας. Ο λόγος που είναι αφιλεγόμενο το εργαλείο αυτό Βέβαια, ο βασικότερος είναι η διαφθορά. Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι η δημοσιονομική στήριξη οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφθορά. Δεν έχουμε αποδεκτικά στοιχεία γι' αυτό. Εάν δούμε το πώς εξελίσσονται τα πράγματα συγκρίνοντας χώρες που έχουν λάβει δημοσιονομική στήριξη ε, στην κόκκινη γραμμή και σε αυτές που δεν έχουν λάβει στην μπλε γραμμή, βλέπετε ότι το θέμα είναι πώς γίνεται αντιληπτή η διαφθορά, πώς μετράτε με, τη, με τα κριτήρια διαφάνεια και καλή διακυβέρνηση ε, που έχει καταρτήσει η Παγκόσμια Τράπεζα. Οι χώρε που έχουν λάβει δημοσιονομική στήριξη τα πήγαν πολύ καλύτερα ω προ τον έλεγχο και την αντιμετώπιση τη διαφθορά από αυτέ που δεν έλαβαν. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει διαφθορά βέβαια, αλλά πολλοί από του υπευθύνου των αξιολογήσεων τείνουν να πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα έχει σχέση περισσότερο με την καλή λειτουργία του όλου συστήματος ούτως ή άλλως που επιτρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια, η θέση του γενικού ελέγκτη, η διακυβέρνηση, η, η εκδίκαση υποθέσεων που φτάνουν πλέον μπροστά στα δικαστήρια και εκδικάζονται πραγματικά. Εάν δούμε τώρα το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής στήριξης στην οικονομική ανάπτυξη, τίνουμε να πιστεύουμε ότι οι χώρες που έχουν λάβει δημοσιονομική στήριξη έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη από τις χώρε που δεν έχουν λάβει. Δεν φαίνεται όμω να υπάρχει άμεσο συσχετισμό μεταξύ καλή διακυβέρνηση και οικονομική ανάπτυξη. Τώρα θα πρέπει να είμαι πολύ σύντομος. Αντίκτυπος δεν υπάρχει ούτε ως προς την ούτε προς τους δείκτες της ανθρώπινης ανάπτυξης του βιωτικού επίπεδου. Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ δημοσιονομικής στήριξης και της ε, αύξησης του πολλαπλασιασμού των πόρων για τον κοινωνικό τομέα, όπως έλεγα, αλλά ως προς το συγκεκριμένο αντίκτυπο. Υπάρχουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία ότι χώρε που έλαβαν δημοσιονομική στήριξη είχαν υψηλότερη οικονομική αύξηση από χώρε που δεν την έλαβαν αλλά χώρες που έλαβαν δημοσιονομική στήριξη επίσης έχουν μεγαλύτερο υψηλότερο λόγο μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και καταπολέμησης της φτώχειας από τις χώρες που δεν πήραν. Θετικό και αυτό. Όμως, χώρες που έλαβαν δημοσιονομική στήριξη, όπως είπα, τα πήγαν καλύτερα ως προς την καταπολέμηση της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη. και στην περίπτωση των δικτών ανθρώπινης ανάπτυξης. Εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα από την ε, Κομισιόν χάρη με συγκεκριμένους δείκτες και επίσης μπορείτε να δείτε ότι οι φτωχότερες ομάδες τα πήγαν καλύτερα με τους πόρους που έλαβαν από τους κοινωνικούς τομείς, στους, στον κοινωνικό τομέα από ότι σε άλλους τομείς. Δηλαδή, οι φτωχότερες χώρες περισσότερο ωφελήθηκαν στον κοινωνικό τομέα και εκεί δαπάνησαν τα χρήματα από ότι σε άλλους. Αυτά θα τα επιδείξω, δεν έχω χρόνο. Τώρα, για τους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης. Οι χώρες που έλαβαν ε, δημοσιονομική στήριξη βελτίωσαν περισσότερο τις επιδόσεις τους εκεί από ό,τι χώρες που δεν έλαβαν. Εδώ, λόγου χάρη, βλέπετε, αν δείτε τα σκούρα τμήματα του διαγράμματος στις στήλες, τα σκούρα τμήματα αντιστοιχούν στην προσφορά της δημοσιονομικής στήριξης. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του δίκτυου ανθρώπινης ανάπτυξης, μάλλον στο δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης, μεταξύ των χωρών που έλαβαν ή δεν έλαβαν δημοσιονομική στήριξη. Και κάποια από αυτά είναι απευθεία αποτέλεσμα του εργαλείου αυτού. Είναι άρα αποτελεσματική η δημοσιονομική στήριξη. Συμπεράσματα τώρα. Κατά πρώτον, η δημοσιονομική στήριξη ήταν ένα καινοτόμο μηχανισμό για την καταπολέμηση τη φτώχεια. Και αυτό απέτησε ανάληψη τη ευθύνη ιδιοποίηση από τι ε, χώρε δικαιούχου. Ταυτόχρονα όμω οι δωρητέ άρχισαν να παρακάμπτουν, να, να μην ε, τηρούν την ε, αρχή ότι η δημοσιονομική στήριξη είναι ένας τρόπος για να επηρεαστεί και να βελτιωθεί η διακυβέρνηση αντί να ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχεια και να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο σε εργαλείο χρηματοδότησης, το χρησιμοποίησαν ως κίνητρο για την βελτίωση της διακυβέρνησης. Αν δούμε τα αποτελέσματα. Δεν είναι πολύ αποτελεσματική η δημοσιονομική στήριξη προς το να κινήσει μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί να επιβάλλει μεταρρυθμιστικές τάσεις εάν αυτό δεν υποστηριχθεί από τις ίδιες τις κυβερνήσεις δικαιούχους. Ωστόσο, ήταν αποτελεσματική η δημοσιονομική στήριξη όταν χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός χρηματοδότηση για την καταπολέμηση τη φτώχεια. Άρα, όλη την προηγούμενη δεκαετία, κοιτάζουμε σε λάθος σημείο ψάχνοντα τα αποτελέσματα που αναζητούμε. Γι' αυτό έχει γίνει τόσο αμφιλεγόμενη η δημοσιονομική στήριξη. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ Και τώρα τα μέλη τη επιτροπή των αν να Προχωρήσουμε περισσότερο σε βάθος για την ε, ε, παρουσίαση αυτή. Κύριε Μπέρμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα με πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εγώ ήμουν εισηγητής στην Επιτροπή Ολέγχου του Προπολογισμού για την ε, δημοσιονομική στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και βεβαίω ε, ασχολήθηκα και με την ε, εκπόνηση τη πολιτική για τα επόμενα 7 χρόνια, γιατί το εργαλείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακριβώ είναι σημαντικό, επειδή επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημοσιονομική στήριξη ακριβώς ως εργαλείο για να ενισχύσουμε τα, την προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα της Ένωσης. Στη δική σας την έκθεση ε, στηρίζεται στεναρά ότι αυτό δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, κάθε άλλο παρά. Η δημοσιονομική στήριξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, λέτε, με αυτόν τον τρόπο, αποτελεσματικά τουλάχιστον. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω ως προς αυτό, γιατί βεβαίως αυτό είναι ιδιαίτερος ε, ανισχυτικό για μένα που είμαι και εισηγητής. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να προτείνω να ακούσουμε κάποιες παρεμβάσεις πρώτα. Ο κύριος Γκάιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ερώτημα μου έχει παρόμοια, πάει στην ίδια κατεύθυνση με το, αυτό που είπε και ο κύριος Μπέρκμαν. Αν έχω καταλάβει καλά, Δυστυχώ δεν μπόρεσα να διαβάσω την ε, μελέτη σας, αλλά είπατε ότι δεν, υπάρχει συγκεκριμένη σχέση μεταξύ δημοσιονομικής στήριξης και βελτίωσης της διακυβέρνησης στις διάφορες χώρες και της ε, διαχείρισης ε, των οικονομικών στις χώρες δικαιούχους, εάν δεν το υποστηρίζουν αυτό και οι κυβερνήσεις. Ε, προφανώς, αυτό είναι κατανοητό και απολύτως λογικό. Αν τώρα εμείς επιβάλλουμε συγκεκριμένα κριτήρια για την δημοσιονομική στήριξη, αν πούμε, ας πούμε ότι θέλουμε να υπάρχουν ε, ανεξάρτητοι ελεγκτές που θα ενημερώνουν το κοινοβούλιο ή αν ε, λέμε ότι στα Υπουργεία των χώρων, των δικαιούχων θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα έντυπα που θα καταγράφονται οι διάφορες ε, κινήσεις οικονομικές. Αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο στη δική σας τη μελέτη ή αυτές ακριβώς είναι οι προϋποθέσεις που θέλετε να υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Επόμενος, Νόιζερ. Ευχαριστώ. Δεν ε, ξέρω ακριβώς τι θα την κάνουμε αυτή τη μελέτη. Υπάρχουν ε, ε, επικριτικά σχόλια, κυρίως από την πλευρά όσων που λένε ότι δεν ελέγχονται τα, οι φόροι και πηγαίνουν σε χώρες που δεν έχουν καμία καλή διακυβέρνηση, που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ αφήνουμε έτσι πολύ χαλαρά τις ε, κυβερνήσεις να διαχειρίζονται τα χρήματα των φορολογουμένων. Εγώ θεωρώ ότι η έκθεση είναι καλή γενικώ. Είπατε ότι το εργαλείο αυτό είναι αποτελεσματικό, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλύτερα εργαλεία μέτρησης για να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η δημοσιονομική στήριξη, ακριβώς ό,τι αφορά τον τομέα της μείωσης της ε, φτώχειας. Εκεί επιτύχαμε τους στόχους της χιλιετίας. Οι πιο φτωχοί πώς επωφελήθηκαν από την δημοσιονομική στήριξη. Και επίσης ένα σημαντικό σημείο στον ελεκτικό μηχανισμό είναι το εξής οι ε, αντιπροσωπείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί εκείνε μπορούν να ελέγξουν επιτόπου αν αυτέ αν αυτές οι προϋποθέσεις που θέτουμε εμεί ω δωρητέ, πληρούνται ή δεν πληρούνται. Εδώ νομίζω λοιπόν ότι τα εργαλεία αυτά είναι τελείω ανομοιογενή, ε, ακόμη και στις ε, ίδιες αντιπροσωπείες δεν είναι απόλυτα σαφέ αν όντω το εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι επιτυχέ ή όχι. Ευχαριστώ. Γιάννη Μούλτερ. Thank you. Ευχαριστώ. Όταν άκουσα το θέμα αυτό της δημοσιονομικής στήριξης, ε, δεν άκουσα κάτι. Ότι για έναν ε, δωρητή είναι πολύ πιο εύκολο να δώσει στήριξη στον προπολογισμό αντί για στήριξη σε πρόγραμμα. Γιατί ε, μπορεί πολύ εύκολα να, δώσεις έναν, να στείλεις έναν λογαριασμό πολλά εκατομμύρια και να τελειώσει με τις υποχρεώσεις του μπορεί να πει ότι α, εγώ δαπάνησα το 0,7 του ΑΕΠ μου ας πούμε στο τάδε σημείο και 0,6 στο τάδε, στην τάδε χώρα. Αλλά όταν πρέπει κανείς να, να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένα project, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί πρέπει να μελετήσει κανείς και την δομή των, προ... των προγραμμάτων κτλ. Και επίσης κάτι άλλο για την δημοσιονομική στήριξη, κυρίως για την Αφρική. Σε κάποιες χώρες οι κυβερνήσεις δαπανούν πολύ σημαντικά ποσά σε στρατιωτικές δαπάνες και στις μυστικές τους υπηρεσίες, δίνοντας στη δημοσιονομική στήριξη αυτό καθίσταται πιο εύκολο για την ίδια την κυβέρνηση δηλαδή να δαπανίσει χρήματα για να διατηρήσει αυτά τα κονδύλια για, τις, ε, την παρακολούθηση του λαού και για τις ε, στατιωτικές της δαπάνες. Αυτό το λάβατε υπόψη σας, έπαιξε κάποιο ρόλο στους ε, λόγους που καταγράψατε. Madame Κυρία Σαργεντίνη, το λόγο. Δύο ερωτήματα το πρώτο για τα συμπεράσματά σας. Θα πρέπει να αντιλήσω το συμπέρασμα ότι λέτε ότι όταν οι χώρες δωρητές χρησιμοποιούν τη δημοσιονομική στήριξη όχι σαν εργαλείο για την εξάλληψη της ένδυας, αλλά ως ένα κίνητρο για καλή διακυβέρνηση για ευκυβερνησία, ως επιβράβευση για μια κυβέρνηση η οποία έχει επιτύχει κάποια μεγαλύτερη ευκυβερνησία, ότι με τον τρόπο αυτό εξαφανίζεται η αποτελεσματικότητα και δεν είναι αποτελεσματικό εργαλείο. Είναι σωστό αυτό. Δεύτερον, όταν μιλάμε για την δημοσιονομική στήριξη από μια Ολλανδική οπτική γωνία ή μια Ευρωπαϊκή οπτική γωνία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαφορά είναι οι περιορισμοί που έχουν να κάνουν με τις πηγές αυτές δωρεών η δημοσιονομική στήριξη και στις κατοχώρες και, στην, για την Ευρωπαϊκή Κομισιόν δεν είναι χρήματα που μπορεί να δαπανίσει κανείς κατά το δοκούν, είναι χρήματα τα οποία υπόκειται σε κάποιες προϋποθέσεις, σε κάποια αρεσιμότητα. Ποιο τμήμα λοιπόν της δημοσιονομικής στήριξης είναι πράγματι δημοσιονομική στήριξη με την έννοια του κ. Μίλτο και πόσον υποστήριξε συγκεκριμένα σχέδια. Η κυρία Ίγκια Ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να μιλήσουμε και για την εναλλακτική λύση που είναι μέσα για συγκεκριμένα σχέδια. Και η δική μου εμπειρία είναι ότι είναι πιο θετικά, πιο αποτελεσματικά τα σχέδια. Ίσως τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε δει να δείχνουν ότι δεν ήταν αρκετά σαφείς οι προϋποθέσεις οι οποίες τέθηκαν για τη δημοσιονομική στήριξη, ότι ήταν πολύ πιο σαφείς αυτές οι προϋποθέσεις για την στήριξη σχεδίων. Και φυσικά δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να χρηματοδοτούμε ε, συμβούλους και όχι κατευθείαν κυβερνήσεις και προϋπολογισμούς. Εντάξει, λέει ο Μπορούμε να ζητήσουμε τώρα να πάρουμε μια απάντηση για όλε αυτές τις ε, ερωτήσεις από εσά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέροντα τα ερωτήματά σας. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο. Αν δείτε τις προηγούμενες αξιολογήσεις, αν δείτε χώρες οι οποίες πήραν δημοσιονομική στήριξη και χώρες που δεν πήραν δημοσιονομική στήριξη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προσδοκούμε πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στην πολιτική των κυβερνήσεων, αν αυτές οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να δώσουν ιδιαίτερη δημοσιότητα στις πολιτικές τους. Πιστεύω ότι οι πολιτική αυτή μπορεί να αποδώσει μόνο αν και οι χορηγοί και οι κυβερνήσεις που είναι αποδέκτες συμφωνούν για τις προτεραιότητες και για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές τις προτεραιότητες. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν δώσετε μόνο στήριξη δημοσιονομική σε χώρες οι οποίες ε, εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό όμως είναι ένα πολιτικό θέμα, μια πολιτική επιλογή. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τίποτα με την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής στήριξης. Το δεύτερο θέμα για το συσχετισμό μεταξύ δημοσιονομικής στήριξης και κυβερνησίας. Υπάρχει ένας μικρός θετικός, μια μικρή θετική συσχέτιση. Και στις περισσότερες αξιολογήσεις είδαμε ότι οι χορηγοί νιώθουν κάπως απογοητευμένοι σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ευκυβερνησίας στις χώρες οι οποίες επωφελούνται από τη δημοσιονομική στήριξη. Υπάρχει όμως σαφώς θετικός, σαφής θετικός αντίκτυπος όταν βλέπουμε τη δημόσια δημοσιονομική διαχείριση, όταν βλέπουμε τα θέματα λογοδοσίας και διαφάνειας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι χορηγοί έχουν ένα πολύ καλό επιχείρημα για να επιμείνουν να υπάρξουν βελτιώσεις στους τομείς αυτούς, γιατί είναι τα λεφτά των χορηγών τα οποία πηγαίνουν στον προϋπολογισμό και εκεί μπορούν να επιμείνουν σε βελτιώσεις σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ συγχρόνως οι κυβερνήσεις που είναι οι αποδέκτριες των πόρων αυτών ενδιαφέρονται και αυτές να βελτιώσουν σε αυτούς τους τομείς την κατάσταση. Επομένως δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν προκύπτουν βελτιώσεις στην ευκυβερνησία, αλλά ιδίω στη λογοδοσία και τη διαφάνεια, στην διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε ευρύτερε μεταρρυθμίσει, γιατί εκεί δεν υπήρξε, σύμφωνα με τη μελέτη μα, ιδιαίτερο αντίκτυπο. Τρίτο ερώτημα. Τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την έκθεση. Αν θέλουμε να καταμετρήσουμε τα αποτελέσματα που επιτέλεσαν για τη μείωση της Είναι σημαντικό καταρχήν να προσπαθήσουμε να καταμετρήσουμε με διαφορετικούς τρόπους τον αντίκτυπο για τη μείωση της ένδυας. Είδαμε τις προηγούμενες αξιολογήσεις που είχαν γίνει και τις προηγούμενες αξιολογήσεις σε σχέση με το στόχο της μείωσης της ένδυας, αλλά προβήκαμε και σε οικονομετρικές αναλύσεις. Είδαμε την φιλολογία σε οικονομικά περιοδικά και άρθρα για τα θέματα αυτά σε σχέση με το πώς η δημοσιονομική στήριξη προσδιορίζει τη μείωση της ένδυας και όπως είπα προηγουμένως είναι μικρός ο αντίκτυπος αλλά είναι σαφής ο αντίκτυπος αυτός. Υπάρχει μια θετική, ένας θετικός συσχετισμός. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για του οποίους δεν είναι αποτελεσματική η δημοσιονομική στήριξη στη μείωση τη ένδυα. Και όταν μιλάμε ένδυα, μιλάμε για ένδυα σε σχέση με το εισόδημα. Αυτό γιατί η δημοσιονομική στήριξη έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο για να αυξηθούν οι δαπάνε σε ορισμένου τομεί. Αλλά όταν δείτε την οικονομική ανάπτυξη για πολλέ χώρε τη Αφρική δεν υπήρξε αντίκτυπο στην ύπεθρο για του ε, αγροτικού πληθυσμού Δεν υπήρξε έμφαση στη βελτίωση των συνδικών στη Γεωργία. Αυτό αλλάζει τώρα. Εντάξει, θα είμαι σύντομο. Σε τελική ανάλυση, λοιπόν, ο αντίκτυπο για τη μείωση της ένδυας προκύπτει κυρίως από τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτε. Είδαμε για τις ε, δαπάνες στο στρατιωτικό τομέα, αλλά το κοιτάξαμε αυτό. Αν δείτε τη σχέση μεταξύ της ε, δημοσιονομική στήριξη και των δαπανών σε διάφορου τομεί είναι κυρίω στον υγειονομικό τομέα, τον τομέα της παιδείας και υπάρχει και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Στον τομέα της άμυνα δεν έχουμε καμία, δεν έχουμε στοιχεία για συσχετισμό μεταξύ δημοσιονομικής στήριξη και αύξησης των στρατιωτικών δαπανών. Μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις όπως η Ουγγάντα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν υπάρχει σαφή, σαφή συσχετισμός μεταξύ δημοσιονομική στήριξη και στρατιωτικών δαπανών. Εντάξει, θα τα αφήσω εδώ αυτά τα πράγματα. Δεν πρόκειται να απαντήσω περισσότερο γιατί με πιέζει ο χρόνο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Επειδή έχουμε την ακρόαση που ακολουθεί, θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να μα πει αν θέλει να κάνει κάποια σύντομη δήλωση για τα θέματα αυτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σούζαν δίλετε από την ΕΦΚΟ την μονάδα για την ε, δημοσιονομική στήριξη, τα δημόσια οικονομικά και τις ε, οικονομικές αναλύσεις της χώρας αποδέκτρες. Θέλω ε, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Συμφωνούμε και εμείς ότι η δημοσιονομική υποστήριξη έχει αναλάβει μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια. Κατανοούμε ότι με μεγαλύτερη δημοσιότητα έρχεται και η περισσότερη, ο περισσότερος έλεγχος για όλα αυτά τα θέματα και η αξιολόγηση που έγινε, αξιολόγηση που έγινε το 2011 μαζί με την έρευνα του ΩΣΑ έδωσε παρόμοια αποτελέσματα με τις προηγούμενες μελέτες. Όλα αυτά καταδεικνύουν για μας ότι η δημοσιονομική στήριξη μπορεί να δώσει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στους κοινωνικούς τομείς, βελτιώνει τη διαχείριση και τη διαφάνεια των δημοσίων οικονομικών και υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις. Αυτά βέβαια για τα οποία φοβόμαστε είναι ότι μπορεί να αυξήσει την διαφθορά ή μπορεί να εμποδίσει την αύξηση του εγχώριου εισοδήματος. Αλλά δεν είχαμε καθόλου ενδείξεις για αυτά τα δύο στοιχεία που ήταν οι φόβοι μας. Παραμένουν όμως κάποιες ε, προκλήσεις και κάποιες δικαιολογημένες επικρίσεις. Αυτό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν το 2011 είναι μια νέα πολιτική η οποία έχει υποστηριχθεί και από τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ξεφύγει η εστίασή μας από τον κύριο στόχο που είναι η μείωση της ένδυας, αλλά συγχρόνως δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ της ευκυβερνησίας και της μείωσης της ένδυας. Οι δύο αυτοί στόχοι αλληλοενισχύονται τουλάχιστον σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Και πιστεύω ότι η ευκυβερνησία μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και ακόμα και σε αξιολογήσεις που έχουν χρονικό οριζόντα μόνο 10 χρόνια, είναι δύσκολο να διαφανεί αυτό από τη δημοσιονομική στήριξη. Από τις τέσσερις αξιολογήσεις εξέρχεται ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι δεν μπορούμε να αγοράσουμε με χρήματα τις μεταρρυθμίσεις, μπορούμε να υποστηρίξουμε απλώ τις μεταρρυθμίσεις όταν υπάρχει κοινή θέληση και ιδιοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων. Μπορούμε απλώς να τις υποστηρίξουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποδεχτούμε και θα πρέπει να κάνουμε σωστή επιλογή των μεταρρυθμίσεων που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιος από το ελεκτικό συνέδριο θέλει να λάβει το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να υπενθυμίσω στα μέλη των δύο επιτροπών αυτό που είχα πει όταν παρουσίασα το κεφάλαιο 7 ή 8 ποιο είναι για τις εξωτερικές δράσεις στην τελευταία ετήσια έκθεσή μας και στην έκθεση EDF. Στο, και στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν και στη σχετική έκθεση υπάρχουν δύο παράγραφοι οι οποίες αφορούν στην δημοσιονομική στήριξη. Και θα θυμάστε ότι Αυτέ οι ε, παραγραφοί είναι ουσιώδους σημασίας ε, για πολλούς λόγους. Ένα από τον οποίων είναι ότι για μα, ως Ελληνικό συνέδριο, είναι αδύνατον να ακολουθήσουμε τον, ε, το δρόμο που παίρνουν τα χρήματα που πηγαίνουν σε τέτοια προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ανισχυτικό για να το πω ευγενικά. Αυτό λοιπόν, το, αυτή την ε, πορεία που ακολουθούν τα κονδύλια δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Δεύτερον, όταν, όταν μιλάτε για δημοσιονομική στήριξη, ε, θα προσπαθήσω να είμαι προσεκτικός όσα από, μιλάτε για αρκετές χώρες για δημοσιονομική στήριξη σε χώρες που, ε, όπου τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε χώρες με Υπουργεία Οικονομικών που τίνουν πάρα πολύ σε διαφθορά και απάτη. Μπορεί να αναφέρεστε στην ε, διεθνή διαφάνεια, στα δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο και θα πρέπει να σας απασχολήσει σοβαρά. Γιατί δαπανάτε τις, τα χρήματα των φορολογουμένων με πολύ χαλαρό τρόπο. Τρίτον, εάν συνδέσετε τη δημοσιονομική στήριξη με τα συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε το αποτέλεσμα είναι ότι στο μέλλον δεν θα δίνεται πολύ μεγάλη δημοσιομική στήριξη. Αυτά αρχικά τα τρία σχόλια που πρέπει να πω, Πρόεδρε, και χαίρομαι που μου δώσατε το λόγο, που δώσατε το λόγο στο ελεκτικό συνέδριο για να θέσει αυτά τα τρία θέματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή μιας ε, συζήτησης που θα συνεχιστεί. Έχουμε και τη μελέτη, θα την αξιολογήσουμε και θα συμμετάσχουμε στο διάλογο ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Θέλω να, ευχαριστήσω τον κύριο Αντουάν Ντεκέμπ για την τόσο καλά τεκμεριωμένη μελέτη του, η οποία πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες που έχουν εκφράσει, έχει εκφράσει το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι εδώ και 50 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρησιμοποιεί την αναπτυξιακή βοήθεια, χωρίς όμως να υπάρχει αποτέλεσμα στο επίπεδο ένδυας. Ήταν αναποτελεσματική λοιπόν η βοήθειά μας το να βρούμε εργαλεία τα οποία θα κάνουν πιο αποτελεσματική αυτή τη βοήθεια όπως η δημοσιονομική στήριξη. Αυτό είναι κάτω κεφαλαιόδες. Και εφόσον εξεφράστηκε από το ελεκτικό συνέδριο και από ορισμένους άλλους ο φόβος ότι η διαφθορά δεν υπήρξαν αυτοί οι φόβοι. ακριβώ. η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι μπορεί να μειωθεί η διαφθορά με αυτή τη δημοσιονομική στήριξη και να υποστηρίξει και την βελτίωση του δίκτυ ανθρώπινης ε, ανάπτυξης. Θέλω λοιπόν κύριε Δεκέμ να σε ευχαριστήσω για την ελπίδα που μας έχετε δώσει για την ανάπτυξη μέσω της δημοσιονομικής στήριξης. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τα μέλη της Επιτροπής ε, ε, να περάσουν στην οικία μας αίθουσα για να συνεχίσουμε την, τη συνεδρίαση μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει Έτσι έχει κλείσει η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Κοντ και ΔΕΒΕ. Μπορώ απλώς να υπογραμμίσω αυτά που είπε η κυρία Ζολή για την αποτελεσματικότητα των μέσων και την ε, καταπολέμηση της ε, διαφθόρας. Αυτό είναι η κύρια μας μέρημνα Θέλουμε τα χρήματα τα οποία δίδονται από τους φορολογούμενους μας να πηγαίνουν πράγματι στους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ja, nach einer kurzen Veränderung. Μετά από... Κυρία Καλλιέντη, εσείς θα... Εσείς θα λάβετε το λόγο, ναι, από την άλλη μεριά. Francesco. Ja, Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Περνούμε στην ακρόαση για το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για το ολοκληρωμένο πλαίσιο ιστορικού ελέγχου. Η συγγήτρια είναι η Ανδρέα Τσέσκοβα. Θα μας κάνει μια μικρή εισαγωγή στο θέμα. Έχουμε πραγματικά εμπειρογνώμονες και από το Ελεκτικό Συνέδριο και από την Κομισιόν. Έχουμε και εξωτερικούς εκπροσώπους, εμπειρογνώμονες ε, παρόντες στην ακρόασή μας. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Το ανέφερε και το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά βεβαίως και το Κοινοβούλιο στη διαδικασία απαλλαγής επίσης αναφέρθηκε σε αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια βεβαίως δεν έχει υπάρξει απόφαση το της ΚΟΝΤ γιατί δεν θεωρούμε ότι το πλαίσιο είναι παρκές ώστε να εγγυηθεί ότι η δήλωση αξιοπιστίας μπορεί να δοθεί. Με βάση λοιπόν αυτό χαιρετίζω με χαρά τις ε, προτάσεις που υπάρχουν ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ιστορικού ελέγχου. Αυτό είναι η δική μας ανησυχία και είναι και το θέμα βεβαίως της σημερινής ακρόασης. Θα να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας. Θα δώσω βεβαίως πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Τσέσκοβα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. κύριε pane Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη χαρά που μπορώ να κάνω την αρχική παρέμβαση σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα του ολοκληρωμένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια του ε, σχεδίου δράσης της Κομισιόν. Εκ πρώτη όψεως αυτό το θέμα φαίνεται να είναι πολύ τεχνικό και βεβαίως ε, πολύ περίπλοκο ε, και όντως είναι αλλά είναι και ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως ανέφερε μόλις και ο Πρόεδρος. Αν θέλουμε να συζητήσουμε για το σχέδιο δράσης της Κομισιόν, τότε υποθέτω ότι θα πρέπει να θέσουμε μια βασική ερώτηση, την οποία θα πρέπει να απαντήσει τούτη η ακρόαση. Γιατί η Κομισιόν δεν έχει λάβει δήλωση εξοπιστίας. Το σχέδιο δράσης απέτυχε, το αρχικό πλαίσιο απέτυχε, έτσι όπως είχε εκπονηθεί. Μήπως απέτυχε η εφαρμογή του, με ποιο τρόπο η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει με το θέμα αυτό στο μέλλον, με ποιο τρόπο η Κομισιόν θέλει να διορθώσει τα πράγματα στο μέλλον. Οπότε από τούτη την α, άποψη περιμένω πολλά από την παρέμβαση του κυρίου Γκρέι, του πρώην Γενικού Διευθυντή του, της, της Υπηρεσίας Ιστορικού Ελέγχου της Κομισιόν, γιατί ήταν και ένας από τους συγγραφείς αυτού του οδικού χάρτη στα, προς την εκπόνηση ενός ε, πλαισίου ιστορικού ελέγχου. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε ο ίδιος να μας πει ποιες ήταν οι αρχικές φιλοδοξίες και ποιο σκοπό έθεσε η Κομισιόν ώστε να μπορέσει να πάρει την θετική αυτή ε, δήλωση αξιοπιστίας. Επίσης θα είναι πολύ ενδιαφέρον να θυμηθούμε ότι κάποιες δράσεις της ε, Κομισιόν που είχαν ε, ε, μπει στο πρώτο σχέδιο δράσης έγιναν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε προβλεφθεί. Και εδώ σας μιλώ για το νέο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού το οποίο περιλαμβάνει και τις βασικές αρχές κοινού ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου, συγγνώμη, καθώς επίσης και την, ε, τις σαφείς δηλώσεις, υποχρεωτικές δηλώσεις από τα ε, εσωτερικά, από τις εσωτερικές υπηρεσίες για τα δηλώσεις αξιοπιστίας ε, από τα, που προκύπτουν από τις υπηρεσίες των κρατών μελών. Ο κύριος Λεβί από το London School of Economics, τον οποίο έχουμε προσκαλέσει, θα μας, καθαρίσει, θα μας ξεκαθαρίσει, ελπίζω, τις ε, προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το πρώτο σχέδιο της Κομισιόν και ποια ήταν τα απορίσματα. Και χαίρομαι που έχουμε ε, εκπροσώπου εδώ και από την ε, Γενική Διεύθυνση ε, Απασχόλησης, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον, το ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης πέτυχε στα δικά της σχέδια. Η σημερινή ακρόαση για το ολοκληρωμένο πλαίσιο ιστορικού ελέγχου σχετίζεται επίσης και με, το, με την απόφαση για την δήλωση αξιοπιστίας για το 2011 η οποία συζητήθηκε στην ε, Ολομέλεια την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Το Κοινοβούλιο έδωσε νέες κατευθυντήρες γραμμές στην ε, Κομισιόν. Οι πρώτες τρεις προτεραιότητες ίσως δημιουργούν τις αρχικές δυνατότητες έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το θέμα με την δήλωση αξιοπιστίας. Η Κομισιόν και μέσω του κυρίου Κραφ, του εκπροσώπου της, έχει τώρα την δυνατότητα να μας παρουσιάσει τις προθέσεις της. Πιστεύω ότι η δήλωση της Κομισιόν είναι πραγματικά ουσιώδους σημασίας. Το, η δήλωση αξιοπιστίας εξακολουθεί να παραμένει βασικός στόχο για την Κομισιόν. Αυτή η δήλωση αξιοπιστίας είναι πραγματικός, ρεαλιστικό στόχο για την Κομισιόν. Υπάρχουν ε, και διαφορετικές προσεγγίσεις βεβαίως. Ε, Αναγενική διεύθυνση η Γενική Διεύθυνση Άγκρη, Ρίτζο, η απασχόληση, η έρευνα θα πρέπει να έχουν μια ενιαία άγουσα έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν κοινά αποτελέσματα. Αυτό θα είναι δυνατόν. Θα είναι δυνατόν να υπάρξει ένα συνδυασμός προσεγγίσεων έτσι ώστε να επιτευθεί η έκδοση αυτού της δήλωσης αξιοπιστίας. η οποία βεβαίως θα έχει να κάνει και με την αποτελεσματικότητα και την απόδοση. Περιμένω λοιπόν από τους εκπροσώπους και του ελεκτικού συνεδρίου, συγκεκριμένα από την κυρία Καλγιουλάιτ, να μας πει δύο πράγματα για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέσω του σχεδίου δράσης να μας πει αν έχουν υπάρξει αποτελέσματα και αν δεν έχουν υπάρξει, γιατί δεν έχουν υπάρξει. Επίσης, υπάρχει εδώ ε, μια διαφορά μεταξύ του κόστους και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και θα μπορούσε κανείς να πει και κάτι για την ανάγκη ύπαρξης μια συμβαστικής λύσης ε, μεταξύ των παραδοσιακών, ε, της παραδοσιακής προσέγγισης για την δήλωση εξοπιστίας για την, ε, και για την, τον καθορισμό των, του κόστους των ελέγχων αυτών. Επίσης, πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την απόδοση και τη σχετική προσέγγιση με βάση την απόδοση και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Ε, φτάνω προς το τέλος. Ε, ελπίζω ε, ότι ο κύριος Μουή, ο πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας των Συνδικών Ελέγχων, θα ασχοληθεί με το θέμα της, της επιβεβαίωσης της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή θεωρώ ότι θα, πρέπει οι πολίτες να πιστεύουν ότι τα ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να προχωρήσουν με τον τρόπο που πρέπει στη διαχείριση των κονδυλίων. Εμάς βεβαίως αυτό στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος. Βεβαίω θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τι δηλώσει αξιοπιστία που εκδίδονται από τα κράτη-μέλη, γιατί και αυτό το σημείο είναι προβληματικό και το είδαμε και το βλέπουμε μάλλον κάθε φορά στην ε, διαδικασία απαλλαγή κάθε χρονιά. Τουλάχιστον το βλέπουμε από τότε που είμαι εγώ στο Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα επίσης ε, στη συζήτηση να ασχοληθούμε και με το θέμα εξέβρεσης νέων προσεγγίσεων, νέων ε, τρόπων ε, επίλυσης του προβλήματος, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και να δώσουμε και στην αποδοτικότητα την σημασία που της αναλογεί. Το θέμα της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας μπορεί να αποτελέσει ένα ορόσημο έτσι ώστε η δήλωση αυτή αξιοπιστίας να μπορέσει να δοθεί και νομίζω ότι και ο πρόεδρος έχει την ίδια άποψη γιατί έχει πει ήδη ότι αυτή η δήλωση αξιοπιστίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και χαίρομαι για, τις, ε, για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια έκθεση η οποία θα μπορέσει να υποστηριχθεί από τότε την Επιτροπή και θα θέσουμε πραγματικά ένα ορόσημο για την απαλλαγή, για τη σχετική διαδικασία απαλλαγής για τις επόμενες χρονιές. Και ελπίζω και οι επόμενες εκλογές να βοηθήσουν τους νέους ευρωβουλευτές να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Συγήτρια. Θα ακούσουμε τώρα τους εμπειρογνώμονες. Καταρχήν ο Brian Gray, ο οποίος ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ε, ε, υπηρεσίας του προπολογισμού στην Κομισιόν και θα μιλήσει και για, τους, ε, για το δικό χάρτη της Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παραμείνετε μέσα στα ωρία των 10 λεπτών κύριε Γκρέι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 10 λεπτά, αλλά έχω να τόσα πολλά. Ήμουνα γενικός ε, διευθυντής για τον εσωτερικό έλεγχο, αλλά ήμουνα προηγουμένω υπεύθυνο για τους έλεγχους στη Γεωργία, για την περιφερειακή πολιτική και στη συνέχεια ενεπλάκη στη σύνταξη του οδικού χάρτη που έχετε ενώπιόν σας. Επομένως έχω μια μακρά πείρα στα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Μπορείτε να με αυγοβολήσετε, να μου πετάξετε κλουβιά αυγά αν θέλετε, αλλά περί αυτού πρόκειται. Αυτά είναι τα θέματα που με απασχόλησαν. Μιλάμε για ένα οδικό χάρτη που πάει πού Κομισιόν είπε ότι θέλει να επιτύχει μια θετική δήλωση αξιοπιστίας, γιατί η Κομισιόν δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Οι ευρωσκεπτικιστές χαίρονται, επιχαίρουν για την έλλειψη θετικού DAS πιστοποιητικού αξιοπιστίας. Επομένως η Κομισιόν πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα αλλά πάντα είναι στην κρίση του ελεκτικού συνεδρίου για το αν θα δώσει το πιστοποιητικό αξιοπιστία ή όχι. Δεν είναι τη Κομισιόν. Η Κομισιόν λοιπόν προσπάθησε να δημιουργήσει ένα οδικό χάρτη για να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν ήθελε να καταδείξει ότι τα συστήματα ελέγχου και οι έλεγχοι που εφαρμόζονται μπορούν να είναι οι καλύτεροι δυνατοί για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ε, ατέλειες κατασταλίες σε ένα επίπεδο πολύ κοντά στο μηδέν. Το πρόβλημα ήταν ότι το ελεκτικό συνεδρίο έλεγε ότι το επίπεδο σφαλμάτων ήταν πολύ ψηλό. Σωστό ήταν αυτό. Οι εμπλεκόμενοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεράνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά τον προπολογισμό. Τότε η Κομισιόν δεν είχε να, να παραθέσει κάποια επιχειρήματα, ιδίω όταν το επίπεδο σφαλμάτων και ε, ατελειών παρέμενε υψηλό. Το ελεκτικό συνέδριο επίσης κατέγραφε τα επίπεδα σφαλμάτων, αλλά δεν μπορούσε να δώσει μια ανάλυση για τα αίτια αυτών των σφαλμάτων, ούτε μπορούσε να προτείνει διορθωτικά μέτρα για την Κομισιόν. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι ουσιαστικά έλεγε το ελεκτικό συνέδριο ότι ο ασθενής έχει υψηλό πυρετό, αλλά δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί γινόταν αυτό. Ένα μονάχα μικρό τμήμα των δαπανών την χάνει διαχείριση από την Κομισιόν, το υπόλοιπο κυρίω από τα κατημέλη, γεωργία, διαρθρωτική πόρη, από τρίτε χώρε, από διεθνεί οργανισμού, από τα Ηνωμένα Έθνη παραδείγματο χάρη, από αποκεντρωμένου φορεί, από εθνικού φορεί. Όλοι αυτοί δαπανούν τα χρήματα και η Κομισιόν του επιστρέφει τα ποσά τα οποία έχουν δαπανίσει. Η Κομισιόν λοιπόν προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι είναι λογικό το επίπεδο σφαλμάτων για αυτούς τους φορείς, αλλά αυτό δεν περνάει μόνο από το χέρι της Κομισιόν, αλλά έχει να κάνει και με όλες αυτές τις διαφορετικές υπηρεσίες. Το Ελεκτικό Συνέδριο έφερε ένα εξαιρετικό έγγραφο που είναι η γνωμοδότηση για τον ενιαίο λογιστικό έλεγχο και μας έδωσε ιδέες για το τι θα πρέπει να επιτύχουμε, να έχουμε συστήματα ελέγχου που εξασφαλίζουν την σωστή ισορροπία μεταξύ της μείωσης των ατασταλιών και ελλείψεων και από τη μια πλευρά και ενός λογικού κόστους από την άλλη πλευρά. Ενεκρίθη αυτό από την Κομισιόν το, 2010, το 2005, 15 Ιουνίου, με στόχο να υπάρξει μια κοινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ελεκτικό Συνέδριο για το ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα μπορούσε να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Στο δεύτερο μισό του 2005 υπήρξαν μακρές συζητήσεις με το Συμβουλίο, υπήρξε μια ομάδα εργασία η οποία δημιουργήθηκε και επίσης τους κόρπους της Κομισιόν για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Καταλήξαμε σε ένα σχέδιο δράση που ενεκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2006 και αφορούσε δύο χρόνια με δύο, διάμεσες, με δύο εκθέσεις πρόοδου και μια έκθεση αντικτύπου που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει να διαβάζετε. Οι στόχοι ήταν πολύ. Καταρχήν υπήρχε ένα γενικό στόχο που μπορείτε να κατανοήσετε, να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για το τι συνέβαινε στην πράξη. Έπρεπε να εξηγήσουμε ότι δεν ήταν πρόβλημα με του λογαριασμού τη Κομισιόν. Οι λογαριασμοί τη Κομισιόν μετά από το 2008 θεωρούνται ότι δίνουν μια ακριβή και σωστή εικόνα των πραγμάτων. Δεν υπήρχαν προβλήματα με τις ε, πληρωμές που γίνονται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Τα προβλήματα όμως ήταν με τις ε, χιλιάδες ε, αιτήσει πλωμών από τους ε, δικαιούχους σε όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν ήταν το πρόβλημα. Υπάρχει έλεγχος για αυτές τις αιτήσει επιστροφής ποσών. Η Κομισιόν είχε ζητήσει από τα κάτι μέλη να κάνουν τα απαραίτητα. Υπήρξε ένα σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε, το οποίο μπορούσε να καλύπτει τις ε, τελικές πληρωμές, γιατί ήταν πολύ πολύ δάπανο να αντιμετωπίσουμε τις ενδιάμεσες πληρωμές. Ο στόχος μας ήταν να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν σωστό. Και υπήρξαν πολλά χρήματα τα οποία ανακτήθηκαν. Περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ήταν οι ανακτήσεις μας. Υπήρχαν σφάλματα τα οποία οδήγησαν σε ανακτήσεις, όχι από τον χρόνο που γίνεται η η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά από προηγούμενα χρόνια. Υπήρξαν λοιπόν ε, και συμπεράσματα για ορισμένα ελεγκτικά πλαίσια, όπω αυτό τη Γεωργία, και το οποίο πήραμε και είπαμε θα το κάνουμε ένα υπόδειγμα για τι άλλε υπηρεσίε. Δεν μπορώ τώρα να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά αυτό το οποίο προέρχεται από το παράδειγμα τη Γεωργία, να βελτιώσουμε το πλαίσιο αυτό σε όλου του άλλου τομεί. Να δημιουργήσουμε καταρχήν μια στρατηγική ελέγχου για όλες τις ε, χορηγήσεις που γίνονται για να μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος. Να ποσοτικοποιήσουμε λοιπόν το ποσοστό σφαλμάτων για να ξέρουμε ποιοι είναι οι τομείς αρρωγής που δημιουργούν προβλήματα και επίσης να στοχεύσουμε καλύτερα αυτούς οι οποίοι ζητούν υψηλότερα ποσά υπομορφή επιστροφών. Κάθε γενική διεύθυνση είχε ένα ε, έγγραφο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει για να καταδείξουν ότι υπήρχε σωστό ελεκτικό πλαίσιο και να καταλήξουν στο ποσοστό σφάλματος. Και είχαμε και προϋποθέσεις για άλλες ε, διαδικασίες ελέγχου. Προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία, να δώσουμε καλύτερες πληροφορίες ώστε να μην προκύπτουν σφάλματα και προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε και κυρώσεις όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Αν υπήρχε λοιπόν πράγματι κάποιο σφάλμα και κάποιος το έκανε και επίτηδες θα μπορούσαν να υπάρχουν διοικητικές ε, κυρώσεις. Μας ενδιαφέρει επίσης, να έχουμε καλύτερη εταιρική σχέση και με τα κάτι μέλη. Αν τα καταφέραν καλά στη Γεωργία, γιατί όχι σε άλλου τομεί. Εργαστήκαμε λοιπόν πολύ σκληρά στον τομέα των διαφορετικών πόρων για να εξασφαλίσουμε ότι τα κρατη μέλη θα είχαν καλύτερα πρότυπα για το λογιστικό έλεγχο. Και εργαστήκαμε με εκατοντάδες φορέων που ήταν αυτέ που τελικά κατέβαλαν χρήματα στον τομέα των διαφορετικών πόρων. Και εδώ τα πράγματα πιστεύω ότι εξακολουθούν να βελτιώνονται. Προσπαθήσαμε να ενθαρρύνουμε τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια να προσέξουν περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δαπάνη των ε, ενωσιακών ποσών στα κράτη-μέλη. Και δημιουργήσαμε και ένα διάλογο με αυτά τα ελεκτικά συνεδρία. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα ολοκληρωμένο ελεκτικό πλαίσιο, έχουμε μία πυραμίδα ελέγχων. Ξεκινάμε με αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά στις διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα γραφεία του ΟΗΕ σε διάφορα μέρη. Μετά έχουμε τα κράτη-μέλη τα οποία ασκούν κάποιους ελέγχους για τις ε, υπηρεσίες αυτές. Μετά η κάθε Γενική Διεύθυνση πράττει τα απαραίτητα για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη κάνουν σωστά το λογιστικό έλεγχο των ε, τμήματων του προπολογισμού που εφαρμόζουν μετά έχουμε την ίδια την Κομισιόν η οποία αναλαμβάνει ευθύνη για την ε, εργασία αυτή στο δικό της ε, έγγραφο που παρουσιάζει το έργο όλων των γενικών διευθύνσεων. Ελπίζουμε ότι αυτό είναι μια πραγματική και σταθερή βάση για το ελεγκτικό συνέδριο για την ετήσια του έκθεση, ώστε τελικά στην κορυφή της πυραμίδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να δώσει την απαραγή στην Κομισιόν. Μπορούμε λοιπόν να παρουσιάσουμε ιδέες, αλλά άμα θέλει κανείς να αλλάξει κάτι θα πρέπει να παρακολουθήσει και το πώς εφαρμόζουμε. Ζητήσαμε λοιπόν από κάθε Γενικό Διευθυντή στην ετήσια έκθεση να παρουσιάσει τι ενέργειέ του για την εφαρμογή του γενικού αυτού ελεκτικού πλαισίου. Ζητήθηκε από κάθε Γενική Διεύθυνση λοιπόν να παρουσιάσει το πλαίσιο αυτού ελέγχου και το ποσοστό σφαλμάτων, ποια είναι τα συστατικά στοιχεία για τη δική τους ε, δήλωση αξιοπιστία και αν υπήρχαν προβλήματα, ποια ήταν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για να μπορέσουν να διορθωθούν τα εσφαλμένα. Και επίση ο κάθε Γενικό Διευθυντή θα πρέπει να δώσει τη δική του προσωπική δήλωση αξιοπιστία σε σχέση με το έργο των δικών του υπηρεσιών. Η αντίδραση του ελεκτικού συνεδρίου ήταν θετική στα περισσότερα θέματα, αλλά τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στα διαφορετικά ταμεία. Τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να αναλάβουν πλήρη πολιτική ευθύνη με εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Δεν υπάρχουν ακόμα ε, κυρώσει Ευρωπαϊκή Ένωση αν οι δικαιούχοι διεκδικούν υπερβολικά ποσά πέραν αυτών που δικαιούνται. Οι εθνικές κρατικές υπηρεσίες των κρατών μελών φυσικά δεν ενδιαφέρονται να είναι υποκείμενα ε, αντικείμενα χειρώσεων. Υπάρχουν σφάλματα σε ό,τι αφορά και στις, ε, στις δημόσιες προμήθειες για τα διαρθρωτικά ταμεία. Και επομένω, εμείς λειτουργούμε σε επίπεδο λεκτών και όχι σε επίπεδο καταβολής χρημάτων. Είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Σε σχέση με το 2005 η έκθεση του 2011 λέει ότι πάνω από 95% των δαπανών δεν περιλαμβάνει σφάλματα. Υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση σε όλε τι υπηρεσίε τη Κομισιόν για τα θέματα αυτά και τα μετά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο παρουσιάζει καλύτερα όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει καλύτερη κατανόηση από όλου του για τα προβλήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα επιληθούν και το σύστημα ελέγχου είναι πιο αποτελεσματικό. Και γιατί δεν έχουμε όμω θετική δήλωση αξιοπιστή υπάρχει μεγάλο χρονικό, μεγάλη χρονική δια, ε, μεταξύ της έγκρισης ενός διορθωτικού μέτρου και του αποτελέσματος που έχει για το ποσοστό σφαλμάτων. Υπάρχουν πολλά σχέδια τα οποία έχουν μακρές προγραμματικές περίοδου. Χρειάζεται να αλλάξει η νοοτροπία και η κουλτούρα στα κράτη-μέλη και αυτό χρειάζεται χρόνος και εν πάση δεν μπορεί να υπάρχει εγγύηση για μια μείωση κάτω από το 2% του ποσοστού ασφάλματος, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ πολύ δάπορο. Η Κομισιόν λοιπόν μπορεί να καταδείξει ότι έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσει αυτό το πλαίσιο ελέγχου και υπάρχει και αυτή η γενική ιδέα ότι η δαπάνη των χρημάτων δεν πρέπει να έχει σαν μόνο αποκλειστικό στόχο να έχει χαμηλό ποσοστό φαλμάτων, αλλά να επιτύχει η πολιτική αυτή και να είναι αποτελεσματική σε σχέση με την εξυπηρέτηση των στόχων που τη έχουν τεθεί. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Γκρέ. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να μπουν όλα αυτά τα ευρήματα σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Να ακούσουμε τώρα τον ε, καθηγητή Λεβί και να προσκαλέσουμε και, τους, ε, και τον εκπρόσωπο από το London School of Economics να καθίσουν εδώ στο πάνελ. Ίσως ο κύριος Γκρέι να μπορούσε απλώς να αλλάξει θέση για να ακούσουμε την παρουσίαση και των υπολείπων. Ζητώ συγγνώμη για την ε, ε, ανησυχία που προκαλώ. Θα μπορούσατε να έλθετε να καθίσετε από εδώ αν θέλετε. over there. Mr. Mr. Welcome. Uh, Καλώς ήρθατε κύριε Μπασιλέη και να σας δώσω και το λόγο βεβαίως κατευθείαν για να ακούσουμε τη δική σας παρουσίαση. you Δεν ξέρω αν μπορείτε τα 15 λεπτά να τα μοιραστείτε. Ποιος θα ξεκινήσει, παρακαλώ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την ακρόαση. Είμαστε πανεπιστημιακοί. Αυτό που έχουμε κάνει λοιπόν εδώ είναι να σας θα παρουσιάσουμε δύο λογιών, πορίσματα σήμερα. Τα πρώτα που έχουν να κάνουν με τη γέννηση του εσωτερικού συστήματος ε, ελέγχου και το άλλο με τις συγκεκριμένες επιπτώσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης στη συνέχεια. Δεν είμαστε πολιτικοί θύνοντες, είμαστε σύμβουλοι και ερευνητές. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την παρουσίαση. Ε, βασιστήκαμε σε πραγματικές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μεταξύ 2007 και 2008 και σε έγγραφα και αρχεία τα οποία φτάνουν ως το 2012. Ο καθηγητής Μπάζιλι μπορεί να μιλήσει περισσότερο για θεωρητικά μοντέλα και πλαίσια αν ενδιαφέρεστε, αλλά θα χρειαστούν μια-δυο μέρες παραπάνω για την ακρόαση για να γίνει αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν όλοι θα το αντέξουν. Ε, θα προτιμούσα εγώ να σας δώσω το γενικότερο τοπίο εντός του οποίου εντάσσονται ενδιαφέρουσες ε, παρατηρήσεις και συστάσεις από την έκθεση Γκάιερ για την απαλλαγή του δημοσιονομικού έτους 2011, οι οποίες απηχούν ακόμη ηχηρά ε, στις, ε, στους περιορισμούς του τι έχει πετύχει ως τώρα το εσωτερικό σύστημα ελέγχου να, πάμε, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και να θυμηθούμε την αρχική, τον αρχικό στόχο τη πρώτη επιτροπή Επιτροπής Μπαρόζο από τον Ιανουάριο του 2005. Ήταν να πετύχει μια θετική δήλωση αξιοπιστία το 2009 το αργότερο. Αυτό ήταν ένα πρωταρχικός σκοπό, αλλά δεν ήταν στο, στην διακατοίκη του ευχαίρεια να το πετύχουν βεβαίω. Ιδίω καθώ δεν τα είχαν ε, πάει καλά και από την πλευρά των δαπανών. Όπω σημειώνει η έκθεση Γκάιερ, τα πράγματα πήγαν χειρότερα τα δύο τελευταία χρόνια παρά καλύτερα. Αυτό ε, είναι κάτι που είναι πηγή ανησυχία βεβαίω. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα θυμάστε ότι το αρχικό πρόβλημα μπορεί να έχει στο συνδυασμό της θετικής ε, δήλωσης εξοπιστίας με το ενιαίο μοντέλο ελέγχου και την μεταρρύθμιση του συστήματο απαλλαγή. Κάτι που θα μπορούσε κανεί να το, να το πει και μια ένα προσωπικό μανιφέστο που ήταν έμπνευση, όπω το είχε ανακοινώσει εδώ στο Κοινοβούλιο από το 2004 ο Επίτροπο Κάλλα. Αυτό ήταν ένα ανέφικτο στόχο. Πρώτα απ' όλα γιατί ο επίτροπο ανέλαβε ως επίτροπο Καταστροφών, ε, όπως περιγράφηκε σε εμάς η θέση που αναλάμβανε τότε και βεβαίω ε, η στήριξη για να κάνει κάτι τέτοιο ήταν ανάλογη και από τον πρόεδρο Μπαρόζο. Ε, υπήρχε λοιπόν η ιδέα τη θετική δήλωση εξοπιστία με το ενιαίο σύστημα ελέγχου. όμω το 2005 με τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου και εσωτερικός ε, αυτό το σύστημα κατέρευσε. Έτσι ο δικό Χάρτη άλλαξε τίτλο και από το προ μια θετική δήλωση εξοπιστία πέρασε σε ένα εσωτερικό, ολοκληρωμένο εσωτερικό σύστημα ελέγχου. Στην έρευνά μας εντοπίσαμε εκείνη την περίοδο κάποια βασικά σημεία, κάποια κομβικά σημεία από τον Ιανουάριο του 2005 και την υιοθέτηση του προγράμματος δράσης για τον οδικό χάρτη μέχρι τον Ιανουάριο του 2006. Πρώτον, η εγκατάλειψη της θετικής δήλωσης αξιοπιστίας από το 2009 προς, ε, υπέρ, ε, όφελος μάλλον του νέου συστήματος. Έπειτα, αυτό που ονόμασα μανιφέστο του Επιτρόπου Κάλλας, έπειτα η αποτυχία να συμφωνήσουν εθνικές δηλώσεις και να υπογράφονται σε υπουργικό επίπεδο Τρίτον, η αποτυχία να πιστεί το ελεγκτικό συνέδριο για τον ορισμό των σφαλμάτων, τη μεθοδολογία των ελέγχων ή του τους συσχετισμούς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, την ε, άρνηση να δημιουργηθεί ένα κοινό σύνολο για την απλούστευση των κανόνων και το σύστημα ελέγχου εντός των ε, υπηρεσιών της Επιτροπής. Αυτό από τότε δεν βελτιώθηκε πολύ. Οπότε αυτό που διαβάζουμε στην έκθεση Γκάιερ δεν θα επαναλάβω τώρα όλα, όλα τα παραθέματα που έχω καταγράψει, απλώς έχουμε κάποιες βασικές παρατηρήσεις που επιβεβαιώνουν αυτά τα τέσσερα σημεία αποτυχίες για τις αιτήσει επισκοπήσεις των κρατών μελών που δεν προσφέρουν καμία προστιθέμενη αξία για την ανάγκη εναρμόνισης ε, πρακτικών και υπηρεσιών σε ό,τι αφορά ιδίως τη διακοπή την αναστολή των πληρωμών, τη μεθοδολογία που ακολουθείται, τις διαφορετικές δηλαδή μεθοδολογίες για τη γεωργία και τη συνοχή πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή αλλά και τη μεθοδολογία του Ελληνικού Συνεδρίου. Τίποτα από αυτά δεν μας εκπλήσει βεβαίως ε, και λόγω της ε, αρχικής ισορροπής που επιδιώχθηκε από τους ε, εμπλεκόμενους φορείς, την Επιτροπή, της Υπηρεσίας της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελληνικό Μάλλον Συνέδριο και τα κράτη-μέλη. Δεν είναι ότι διαφωνούμε με τον απότερο στόχο μιας θετικής δήλωσης αξιοπιστίας. Είναι κάτι το πολύ αξιέπαινο ως στόχος. Όμως, ενώ όλοι κάτι θέλανε να πετύχει από όλη αυτή την πρωτοβουλία, δεν νομίζω ότι ακριβώς είχαν τον ίδιο στόχο μεταξύ τους. Και κανένα φορέας ή σύνολο φορέων δεν είχε αρκετά πλεονεκτήματα στα χέρια του, περισσότερα από τους άλλους, ώστε να πετύχει ακριβώς αυτό που ήθελε. Στην περίπτωση της Επιτροπής Λόγου Χάρη μπορούμε να πούμε ότι παρά τις ελλείψεις και τις αποτυχίες που εντοπίσαμε, οι υπάλληλοι εργάστηκαν δημιουργικά και εσωτερικός και εξωτερικός με ε, νομικά εργαλεία, όπως τους νέους δημοσιονομικούς ε, κανονισμούς, το πολυ πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, του νέου κανονισμού για τα διαφορετικά ταμεία κλπ. Και νέε μορφέ διοργάνωσης που είχαν δημιουργήσει οι εκθέσει διαχείρισης κοινοπρόντι. Ε, το CFS, το IES, το AR. για να προχωρήσουν οι προτεραιότητε. Είναι πολλά λοιπόν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να γίνουν και ήταν και μεγάλη δυσκολία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επηρεάσει τα κράτη-μέλη. Παρόλο λοιπόν που ήταν περιορισμένος αντίκτυπο, δεν ήταν αμεληταίος. Έτσι, η ε, επιρροή του περιθωρίου αλλαγών αποδείχθηκε πολύ σημαντική για την πραγματική μεταβολή του συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου στην Γενική Διευθύνση Απασχόλησης ιδίως. Έκανε πολύ συγκεκριμένα σχόλια έκθεση Γκάιερ και για άλλες γενικές διευθύνσεις όπως για τις Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας και Περιφερειών και δεν είναι ότι είναι μια ε, εξαίρεση η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Πάντως η έκθεση εκφράζει την ε, ικανοποίησή της που το ποσοστό σφάλματος είναι πολύ κοντά στο αποδεκτό όριο. Είναι κάτι σαν να λέει, ε, σαν να δίνει εύσημα στην Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Όμως μιλάμε για μια γενική διεύθυνση με σοβαρά προβλήματα και ποσοστά σφάλματος όπως είχε εντοπίσει το ελληνικό συνέδριο στην μέση της δεκαετίας του 2000. Υπήρξε μεγάλη πίεση από το 2007 και μετά για να βελτιώσει τις επιδόσεις της αυτή η Γενική Διεύθυνση. Όπως θα ξέρετε, ε, το νομοθετικό κεντρικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας βελτίωσης ήταν ε, ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός που έδωσε στις Γενικές Διευθύνσεις Απασχόλησης και Περιφερειών νέες αρμοδιότητες για να μπορούν να διακόψουν πληρωμές και να επιβάλλουν νέα εποπτεία για τις υποχρεώσεις ε, συμμόρφωσης του εκτελεστικού φορεί των κρατών μελών. Νέα εργαλεία λοιπόν και πρακτικέ που συμπεριλάμβαναν την αυτοματοποίηση τη ενεργοποίηση τη διακοπή των πληρωμών, ε, την επιβολή ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων τρίμηνιαίου και πιο εντατικού, την de facto ε, αναπομπή της απόφασης ε, αναστολής ή διακοπής στους ε, διευθυντές των geodesk όπως ονομάζονται και την αναβάθμιση της δυνατότητας εσωτερικού ελέγχου που διαχωρίστηκε από τις ερμουδιότητες αποξιολόγησης. Ένα, πλάνο δράσης, ένα σχέδιο δράσης λοιπόν και ένα νέο, ένας νέος μορφότυπος που ε, επιβλήθηκε ε, έξωθεν στην Γενική Διεύθυνση, αλλά και η ανάγκη να επαναοριστεί το ποσοστό σφάλματο, ώστε να υπάρξουν καλύτερε επιδόσει. Τώρα, γιατί η Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, γιατί ήταν αυτή πιο πετυχημένη τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε υπονοούν ότι εκεί ένα σύνολο φορέων και εμπλεκομένων θεώρησαν ότι δέχονται επίθεση από πολλές διαφορετικές πλευρές και ότι ουσιαστικά βρίσκονται σε ένα άφυλο περιβάλλον. Στη Γενική Διεύθυνση για πολλά χρόνια είχε κρατήσει μια τέτοια κατάσταση που οδήγησε σε μια τέτοια νοοτροπία. Γι' αυτό και υπήρξαν κίνητρα για δράση. Ένα κλίμα φόβου και απειλής ήταν η βασική αιτία για τις αλλαγές της αποφάσεως. Αλλά και το γενικότερο τοπίο που επέτρεψε να εξευρεθούν λύσεις. Αυτό είχε να κάνει βέβαια και με το πόσο μπορούσαν να ακολουθούν τις, προδιαγραφε... τις γραφειοκρατικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζονται στους κανόνες ή την ε, άποψη για τα κράτη-μέλη που συνήθως θεωρούνταν υπεύθυνα για τα ποσοστά σφάλματος και για τα ίδια τα σφάλματα. Η επιτάχυνση βέβαια έγινε με τον τίτλο 6 και με το απερχόμενο ε, σύστημα, το σύστημα που σιγά σιγά καταργήθηκε. Τώρα από πού προέρχονταν οι απειλές. οι προφανής ήταν η ετήσια έκθεση αξιοπιστίας, το ποσοστό σφάλματος, η ετήσια απαλλαγή από, το, από την Αρμόδια Κοινοπολιτική Επιτροπή, οι απόψεις των ίδιων των επιτρόπων και του σώματος των επιτρόπων, Επίσης ε, τα όσα δήλωναν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως η Όλαφ. Εδώ έπρεπε να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου και βεβαίως μέχρι τότε η Γενική Διεύθυνση ε, Απασχόλησης βρισκόταν στο λάθος σημείο μιας σχέσης έλλειψης ισορροπίας. Έπρεπε λοιπόν να βρει στρατηγικές για να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές, να τις αναχαιτήσει, χωρίς όμως να επιδεινώσει τις σχέσεις με τους άλλους φορείς και να αντλήσει ε, ωφέλη. Γι' αυτό γενικώ προτιμήθηκε η ρυθμιστική προσέγγιση με στοχοθέτηση του συστήματος υποχρεώσεων συμμόρφωσης των κρατών μελών και των συστημάτων τους η νέα, το νέο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να πιέζονται τα κρατημέλη ήταν η διακοπή των πληρωμών. Από άποψη γραφειοκρατική αυτή η αυτοματοποίηση των νέων κυρώσεων ήταν ε, κάτι το επιθυμητό, διότι έδινε τη δυνατότητα να προβάλλονται αξιώσει για συγκεκριμένα προγράμματα που ενδεχομένω να είχαν επιλεγεί αυθαίρετα από του ε, διευθυντέ των Geodesks. Ε, αυτό ήταν κάτι που δυσκόλευε τα περισσότερα κράτη-μέλη. Όμω έτσι μεταφέρθηκε η απειλή από, τα, από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση στα κράτη-μέλη και στου εκτελεστικού του ε, φορεί. Οι νέε αρμοδιότητε των ε, ε, διευθυντών των εθνικών γραφείων ήταν κάτι που επέτρεψε και η μεταρρύθμιση Κίνοκ πρώτη και υπήρξε έτσι μια ανανέωση των όσων ήθελε να πετύχει και το ΑΕΣ και με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, ε, η αντίληψη για το ποσοστό σφάλματος ήταν κάτι που συνείδευε και με, με τη διάθεση της, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να περιορίσει τα επιτόκια, ώστε να ε, οριοθετήσει καλύτερα το χώρο δράσης της. Εδώ η χρήση του συστήματος διακοπής πληρωμών ήταν σαφές. Είναι δυσκολότερο να πάρει κανείς χρήματα ή να ή μπορεί πολύ πιο εύκολα να διακοπεί η ροή. Το λέει και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. 20% των ποσών ε, το 2009 εκτελέστηκαν ε, και ούτω καθεξής για τις επόμενες χρονιές. Ε, η δυσκολία είναι τα προγράμματα λοιπόν και να επιλεγούν και να λειτουργήσουν. σε full ταχύτητα. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση και την εφαρμογή των προγραμμάτων θα μπορούσε να είναι ένα αποδεκτό τίμημα για την συμμόρφωση όμως. Αυτός ο κατάλογος προτεραιοτήτων φαίνεται να έχει εξελιχθεί. Η έκθεση Γκάγερ κάνει λόγο και για τις επιδόσεις ε, των ελέγχων, των οποίων η μέτρηση έχει γίνει πιο σημαντική από την επιδίωξη των ίδιων των στόχων. Βεβαίω, έναν ιδανικό κόσμο, η τέλεια συμμόρφωση και οι τέλειε επιδόσει είναι, κάποια, είναι πράγματα που μεταξύ του μπορεί να μην είναι ασύμβατα. Όμω, στον, πραγματική, στον πραγματικό πολιτικό χώρο, στην αρένα, την πολιτική, ε, πάντοτε πρέπει να υπάρξουν ε, ανταλλάγματα για να επιτύχει κανεί το ένα ή το άλλο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω. Τι είναι πιο σημαντικό, καλύτερε επιδόσει ή καλύτερη συμμόρφωση. Ευχαριστώ. We Ευχαριστώ. Ε, στις 6.30 όμως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Στις 6.30 ακριβώς, οπότε πρέπει να πάρουν όλοι το λόγο. Γι' αυτό θα σας ζητήσω να είσαστε παρακαλώ σύντομος. Είπα 15 λεπτά και τώρα ε, τα έχουμε περάσει ήδη. Ξεκινήσατε στις ε, 4.30 think uh, Ίσως ε, να υπάρχει χρόνος να υπάρξουν έτσι μια, να μια ανταλλαγή απόψεων και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα πω όμως δύο πράγματα. Το πρόγραμμα λέει ότι ένα από τα ερωτήματα είναι ότι η ε, τη απουσία μη α, α, θετικής α, αξιοπιστίας τι σημαίνει ότι το πρόγραμμα ε, απέτυχε. Μπορούμε να το αναλύσουμε με πολλούς τρόπους αυτό, αλλά η δική μου απάντηση είναι ε, σαφώς όχι. Ένας λόγος για την αρνητική αυτή απάντηση που δίνω είναι ότι το IICF, το ολοκληρωμένο πλαίσιο ιστορικού ελέγχου, δεν ε, ε, δημιουργήθηκε ουσιαστικά για αυτό το στόχο παρόλο που ο, το, ο στόχος για να υπάρξει μάλλον, το να υπάρξει μια θετική δήλωση εξοπιστίας ήταν το κίνητρο αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δυνατοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να αναλάβει διαχειριστικά καθήκοντα για τον τρόπο με τον οποίο θα οι, προγραμμα... οι και για τον τρόπο με τον οποίο ε, εκτελούνται τα προγράμματα. Και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο σοβαρό. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν λαθασμένο να αξιολογήσουμε το ολοκληρωμένο πλαίσιο ιστορικού ελέγχου μόνο επί τη βάση του αν δόθηκε θετική δήλωση αξιοπιστίας. Στα αρχικά σχόλια της εισηγήτριας εγκάθισαν δύο ερωτήματα. Ένα ήταν ε, κατά πόσο υπήρξε κακό σχεδιασμός και νομίζω ότι αυτό χρειάζεται μια ε, διτή απάντηση. Νομίζω ότι αυτό που είδατε εσείς είναι ότι οι στόχοι η προσέγγιση της δημοσιονομικής εποπτείας που ελήφθη από το ελεγκτικό συνέδριο μεγεθύνθηκε μέσω όλων των αναδιαρθρώσεων που έγιναν στα συστήματα συμμόρφωσης και ελέγχου. Οπότε πρέπει να επιστρέψουμε στο ερώτημα αν είναι σωστά ε, σχεδιασμένη η δήλωση αξιοπιστίας, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι μεγέθυνση της δήλωσης αξιοπιστίας ως ε, βασικό πρόγραμμα και ως βασική πολιτική. Ένα άλλο ερώτημα που έθεσε η συγκήτρια είναι το αν ε, εφαρμόστηκε επιτυχώς ή όχι. Αυτό που είπε ο, ο καθηγητής Λεβί είναι ναι, Ξεχωρίζουμε βέβαια το θέμα αυτό από το αν ήταν καλό ο σχεδιασμό του. Ο σχεδιασμό και η εφαρμογή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το θέμα είναι το πώ θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό εμεί στο LSE είναι ότι θα το χρησιμοποιήσουμε θετικά, ω δηλαδή μια περίπτωση θετική ε, έκβαση. Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε για το σχεδιασμό, υπήρξε, υπήρξαν πραγματικά ε, σημαντικές ε, ε, εμπνεύσεις σε ό,τι αφορά την πρακτική που ειδικά το σύστημα ολοκληρωμένου ιστορικού ελέγχου θα μπορέσουν να το καταστήσουν λειτουργικό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το θέμα είναι αν ήταν τελικά δυνατό να αλλάξει το σκεπτικό από το να υπάρχει ένα επταετές πρόγραμμα στο να περάσουμε σε ένα εφταετές πρόγραμμα με ετήσια αξιολόγηση. Αυτό ήταν το μεγάλο βήμα που έγινε, αυτό ήταν το άλμα που έκαναν και νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ε, διαδικασίες ε, έτσι ώστε να γίνει αυτή η μετάβαση και νομίζω ότι πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η ε, επιλογή της πολιτικής και η εφαρμογή του προγράμματος. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Να ακούσουμε κάποιες σύντομες ερωτήσεις τώρα. Ποιο θα πάρει πρώτο το λόγο, η συγκίτρια, κυρία Τσέσκοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ, εγώ δεν θέλω να αφήσουμε τα διαφορετικά ταμεία απ' έξω από αυτή τη συζήτηση, αλλά προς το παρόν θα σταθώ σε ορισμένα θέματα τα οποία ήθελα να θέσω για μένα. Η έλλειψη κυρώσεων είναι ένα κομβικό θέμα. Το θέμα των δημοσίων προμηθειών και του τρόπου με τον οποίο Τονται όλες αυτές οι συμβάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το προγραμματικό διάστημα 2007-2013 υπήρξε μια βελτίωση, αλλά για την αξιοπιστία δεν έχει υπάρξει πραγματικός αντίκτυπο στα θέματα αυτά. Δεν έχουμε καταλήξει σε ένα θετικό πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Οι αναθεωρημένοι κανόνες είναι πιο λυσιτελείς βέβαια, αλλά το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 να αποδώσουν κάποιους καρπούς. Είπατε ότι υπάρχει αν, ανίσ έλλειψη αντιστοιχίας, μια αναντιστοιχία μεταξύ των ε, νέων κανόνων και, των, ε, και της μείωσης των ε, σφαλμάτων. Το ελεκτικό συνέδριο θέλει από τη μια μεριά να μειώσει τα σφάλματα, Από την άλλη πλευρά όμως θα να εξασφαλίσει και την ανάκτηση των ποσών τα έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. Και υπήρξαν επίσης και προσπάθειες να εξασφαλιστούν εξοικονομήσεις στις ελεγκτικές διαδικασίες. Όλα αυτά έχουν επιρροή στην επίτευξη του, πιστοποιητικού, του θετικού πιστοποιητικού αξιοπιστίας. Είναι λοιπόν κατά την άποψή σας εφικτό το να φτάσουμε σε αυτό το, το πιστοποιητικό αξιοπιστίας το οποίο είναι θετικό ή κάτω από τις σημερινές συνθήκες είναι κάτι το αδιανόητο. Και ποιες είναι οι ε, διαδικασίες που πρέπει να τροποποιηθούν κατά την άποψή σας από την Κομισιόν, αν πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση το ελεκτικό συνέδριο, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα για μένα. Και εν τέλει, ποια είναι η άποψή σας για την ε, στάση που κρατούν τα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά. Τι θα έπρεπε να κάνουν τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουν ότι μπορεί να προκύψει ένα σωστό έλεγχο των μέσων των κοντιλίων τα οποία δίδονται. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο θέλει να λάβει το λόγο. Σα παρακαλώ λοιπόν να απαντήσετε με ποια σειρά τώρα. Εγώ διστάζω εδώ να απαντήσω γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης για να σας δώσω κάποιες ιδέες για το τι έγινε για να μειωθεί το ποσοστό σφαλμάτων θα πρέπει να εξασφαλίσει κανείς ότι στο τοπικό επίπεδο, στους δήμους, στις ε, κοινότητες, στις περιφέρειες, αυτοί οι οποίοι κάνουν την τελική καταβολή των ε, ποσών, θα πρέπει να έχουν επίγνωση, απόλυτη επίγνωση της σημασίας της, ε, του εντοπισμού των σφαλμάτων και της διόρθωσης, γιατί η Κομισιόν εργάζεται μονάχα σε ένα υπερκείμενο επίπεδο, σε ένα πιο ψηλό επίπεδο για όλα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο κάθε δήμος, η τελευταία κοινότητα, όσοι εφαρμόζουν αυτά τα μέσα και τα κονδύλια, θα πρέπει να γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι αυτά. Είναι πολύ δύσκολο θα γίνει αυτό πραγματικότητα. Αλλά η Κομισιόν τουλάχιστον μπορεί να εξασφαλίσει ότι όταν κάτι πηγαίνει στραβά και διαπιστώνεται, τα κρατη αναλαμβάνουν κάποια διορθωτική δράση και αν τα κρατη δεν αναλαμβάνουν διορθωτική δράση, τότε η Κομισιόν πρέπει να αναστείλει την καταβολή αρρωγών το οποίο τα κρατη φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Μέχρι ότου η Κομισιόν είναι ικανοποιημένη ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό, αλλά τελικά υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς και άτομα τα οποία διαχειρίζονται το σύστημα σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο τώρα. Πιστεύω ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιώσουμε την, ε, την απόδοση των κρατών μελών είναι φυσικά να σταματήσουμε να τους δίνουμε χρήματα και επομένως η αναστολή προγραμμάτων και χορηγήσεων μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Αυτό καταδεικνύεται και από ορισμένα στοιχεία της Γενικής Διεθνής Απασχόλησης. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι με τον τρόπο αυτό καθυστερεί η εφαρμογή προγραμμάτων και ε, ουσιαστικά δημιουργεί παρεμβολές με άλλους στόχους που έχει θεσπίσει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να βελτιώσουμε τις οικονομικές συνθήκες στα κράτη-μέλη και να έχουμε καλύτερη εφαρμογή προγραμμάτων σε αυτούς τους τομείς. Είναι δύσκολη απόφαση λοιπόν να ληφθεί το να αναστείλει κανείς τα κονδύλια αυτά, να ζητήσουμε απόλυτη συμμόρφωση, ακόμα και αν αυτό θα σημαίνει μεγαλύτερη ε, δυσκολία στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Μήπως αντίθετα θέλουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διευκόλυνση των προγραμμάτων αρρωγής ώστε να μην υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες οι φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα να υποπέσουν σε σφάλματα. Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει και ένα πιο χαλαρό πλαίσιο ελέγχου. Αυτή η συζήτηση γίνεται από ό,τι ξέρω για τα διαδοτικά ταμεία τα τελευταία 30 χρόνια και δεν βλέπω να έχει υπάρξει μια έκβαση υπέρ της μιας ή τη άλλη άποψη και ούτε στα επόμενα 30 χρόνια είναι πιθανό να λυθεί αυτό το δίλημα. Ευχαριστώ. Ποιο θέλει να το λόγο? Για το ερώτημα του αν θεωρείτε ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί ένα θετικό ντάς, ένα θετικό πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, αλλά μπορώ να θέσω το ερώτημα αν ευσταθεί αυτό το ερώτημα, γιατί εδώ βρισκόμαστε σε ένα χώρο όπου μια ουσιαστική αξιολόγηση των διοικητικών προγραμμάτων θα ήταν απαραίτητη και να γίνει μια αξιολόγηση στον τομέα αυτό. Εκεί μπορεί να θέσει το ερώτημα του κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και κάτι ακόμα που συνδέεται με όλα αυτά είναι ότι όπως σας εξηγούσα προηγουμένως μπορείτε να θέσετε το ερώτημα του γιατί υπάρχει αυτό το κατόφλιο του 2% σε ό,τι αφορά την ε, απουσία σφαλμάτων και από πού προέρχεται. Γιατί αν δώσουμε ειδική σημασία στο 2% θα πρέπει να ξέρουμε γιατί το 2% και όχι κάποιο άλλο ποσοστό. Δεν είμαι λογιστής, ο κύριος Γκρέι ίσως γνωρίζει περισσότερα για τα θέματα αυτά από μένα, αλλά μου λένε ότι για το επάγγελμα των λογιστών το 2% ήταν μια καλή πρακτική για την παρουσίαση ισολογισμών ενός των λογαριασμών κάποιας οντότητας, κάποιας επιχείρησης και δεν πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ ενός ισολογισμού μιας επιχείρησης και ενός λογιστικού ελέγχου για την νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών που συνδέονται με τα κοινοτικά προγράμματα. Αλλά έχουμε δύο διαφορετικά αντικείμενα σε αυτήν την περίπτωση και μπορεί ενδεχομένω να θέλετε να επανέλθετε σε αυτή την αρχή μετά από την έγκριση της συνθήκης της Μαστρίχτης. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει ενδεχομένω να θέσουμε γιατί είναι μια ιερή αγελάδα αυτό το 2% για όλους. και ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν να κάνουμε μια εκ του μηδενός επαναξιολόγηση των προγραμμάτων για το πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται με αυτόνομο χαρακτήρα από το ελεκτικό συνέδριο και ενδεχομένως θα πρέπει και τα άλλα θεσμικά όργανα να ενδιαφερθούν και να συμβάλλουν στο, στην προβληματική αυτή. Όπως είπα προηγουμένως, η Κομισιόν έχει ουσιαστικά με τη δράση της μεγεθύνει την ε, επίπτωση της τάσης του ελεκτικού συνεδρίου για τα θέματα αυτό. Και αν θέλετε να δείτε τις ε, πρακτικές οι οποίες γίνονται και οι οποίες είναι ουσιαστικά αλληλένδετες, ίσως θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το κατόφλιο του 2% όταν εφαρμόζεται σε κάθε είδους προγράμματα, και όχι μονάχα σε προγράμματα όπου η Κομισιόν ελέγχει τις δικές της δαπάνε και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ίσως να είναι ενδιαφέρον να το αντιμετωπίσουμε. Εντάξει. Πλησιάζουμε λίγο πιο κοντά στον πυρήνα του θέματος και συνήθως αυτό σημαίνει ότι θα προκύψουν και άλλα ερωτήματα για τα θέματα αυτά. Ίσως όμως είναι καλύτερο να προχωρήσουμε με την ημέρησια διάταξή μας και μπορείτε ίσως να λάβετε μέρος και στη δεύτερη συζήτηση, αλλά προς το παρόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Μάνφερτ Κράφτ, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής για τον προϋπολογισμό και ίσως θα μπορέσουν να προκύψουν και κάποια ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε εσά. Είστε αναπληρωτής, Γενικός Διευθυντής της Γενικής ε, ε, Διεύθυνσης και ο τίτλος του, της παρουσίασής του είναι αν είναι ρεαλιστικός στόχος, αν είναι το ιερό δισκοπότηρο το θετικό πιστοποιητικό αξιοπιστίας και κατά πόσον υπάρχουν ορθολογικές και πρακτικές λύσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ίσως ο τίτλος λοιπόν δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μετά η κυρία Κάρστη Καλλιουλάντ θα λάβει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και θα ήθελα και για τους δύο να σας, να σας παρακαλέσω να σε 10 λεπτά και μόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο για να παρουσιάσω τη θέση της Κομισιόν και την σε σχέση με τις ε, θετικές δηλώσεις ε, αξιοπιστίας, ε, ευχαριστώ που αναφέρετε και εσείς το ιερό δισκοπότερο, γιατί καθιστά σαφέ ότι μιλούμε για κάτι που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και ακόμη και αν το έχει κανείς μέσα στα χέρια του μπορεί πολύ εύκολα να το χάσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα, πρέπει, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Επίσης, μιλήσατε για τα 2.000 χρόνια για τα οποία ψάχνουμε για το ιεροδισκοπότηρο. Εδώ και 18 χρόνια ψάχνουμε για την θετική δήλωση αξιοπιστίας. Η Κομισιόν τουλάχιστον ψάχνει. Είναι ρεαλιστικό λοιπόν αυτή η αναζήτησή μας. Στην δική μου παρουσίαση θα ήθελα καταρχάς να σας αναφέρω ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση. Οι προηγούμενοι ομιλητές ήδη μίλησαν σχετικά για αυτή και θα ήθελα να σας εξηγήσω τι δεν έχει πάει καλά και τι μπορεί να γίνει στο χρόνο που έχω βέβαια στη διάθεσή μου δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Θα επικεντρωθώ μονάχα σε κάποια σημεία κλειδιά για, τις, για τους οδηγικούς ε, παράγοντες που όντως κάνουν τη διαφορά και θέλω να μιλήσω επίσης για την ε, μεικτή διαχείριση που επίσης βρίσκεται στον πυρήνα του ολοκληρωμένου πλαισίου ιστορικού ελέγχου και το οποίο βεβαίως ε, λαμβάνει περίπου πάνω από το 80% του προπολογισμού. Και τέλος, δεν θα παραλάβω αυτά που είπε ο Brian, ο Michael και ο Roger, συμμερίζομαι πολλά από αυτά που είπανε. Ξεκινώντας λοιπόν να πω ότι αν το ολοκληρωμένο πλαίσιο ιστορικού έλεγχου ήταν επιτυχία, ε, ε αναφαντών σας λέω ναι, ε, πρέπει, και μπορώ να σας το αποδείξω χρησιμοποιώντας μονάχα πληροφορίες που προέρχονται από έγγραφα τα οποία αναφέρθηκαν από τον Brian. Όλες αυτές οι πληροφορίες που χρησιμοποιώ στην παρουσίασή μου προκύπτουν από τις ε, τήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων που υπογράφονται από τους Γενικούς Διευθυντές της Κομισιόν, προκύπτουν από τις ε, συνθετικές εκθέσεις που υιοθετήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο από την Κομισιόν και επίσης θα αναφερθώ και στο σημείο 6 των λογαριασμών, το οποίο στο δικό μου επίπεδο εγκρίθηκε και βεβαίως αργότερα από την Κομισιόν στο σύνολό της. Δόθηκε σαφής απάντηση ήδη σε σχέση με τους πολιτικούς στόχους. Ο πολιτική, οι πολιτικοί στόχοι εξακολουθούν να είναι να ε, επιτευχθεί ε, η θετική δήλωση εξοπιστία. Το αναφέρει η έκθεση Γκάιερ, το αναφέρουν οι συστάσει τη Κομισιόν. Το καθιστούν επίση απολύτω σαφέ και αναφέρεται σαφώ και η δέσμευση τη Κομισιόν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Πάρα πολύ συγκεκριμένε λοιπόν οι αναφορέ σε σχέση με τα όσα είχαμε δει στην διαδικασία απαλλαγή του 2011. Αλλά αν δείτε τι διάφορε γενικέ διευθύνσει, όντω υπάρχουν κάποιε αποχρώσει. Για παράδειγμα, η συνοχή ο Επίτροπος Χάν σαφέστατα είπε ότι θα επιτύχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό λάθους στο στιγμή του κλεισίματος, κάτω του 2%. Όταν δηλαδή έχουν παρέμβει όλοι οι διορθωτικοί μηχανισμοί και έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να δώσουν αποτελέσματα. Ταυτόχρονα η κυρία Γκίγεν Κεν είπε ότι μάλλον θα είναι δύσκολο να υπάρχει ε, πίπεδο λάθους κάτω από 2%. Γιατί ακριβώς λόγω των αποτρεπτικών, του αποτρεπτικού κόστους που συνδέεται με την επίτευξη αυτού του στόχου. Για παράδειγμα, στο τέλος κανένας δεν θα μπορεί να ζητήσει κοινωτικά κορδίλια πια, λόγω ακριβώς της ε, κριτικής που, ε, υπάρχει και λόγω της, ε, του ότι δεν δίνεται έμφαση στην αποδοτικότητα και, ότι, και επειδή οι διατάξεις είναι πολύ αυστηρές. Ποια είναι λοιπόν η τρέχουσα κατάσταση. Για τους λογαριασμούς, Έχουμε σαφείς ε, εκθέσεις από το 2007, όχι αποτύχει, αλλά επειδή έχει γίνει τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Ε, ο εξυγχρονισμός δηλαδή των λογαριασμών. Μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να μην χάσουμε το ιερό δισκοπότηρο. Να μην χάσουμε δηλαδή ε, το εξή, ότι η Δημοσιονομική Αρχή, ο νομοθέτης και τα κρατημέλη θα λειτουργήσουν σε ό,τι αφορά τα ε, μετρητά. Έχουν λογική χρήση μετρητών. Ακόμα λοιπόν εκεί υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, αλλά θεωρούμε ότι τους έχουμε υποέλεγχο. Βεβαίως κάποιες φορές μπορεί να υπάρξουν και πλήξεις. Τώρα, πάμε στις ε, ε, συναλλαγές ε, στις οποίες βασίζονται οι ευρωπαϊκοί λογαριασμοί. Εκεί υπάρχουν μικτές, είναι μικρά τα στοιχεία. Το ιερό δισκοπότηρο λοιπόν στα πλαίσια του DAS δεν είναι το ίδιο με το ιερό δισκοπότηρο από μόνο του. Το ιερό δισκοπότηρο είναι ένα πράγμα. Το DAS, η θετική δήλωση αξιοπιστία, παρατηρίζεται από πολλά από πολλέ πτυχές. Ας πούμε για τα έσοδα. Έχουμε θετική ε, γνωμοδότηση. Ο, το ποσοστό λαθού στην τελική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ήταν 0,8%, δηλαδή κάτω από το όριο σημαντικότητα. Για τι ε, δαπάνε έχουμε επίση θετική ε, γνωμοδότηση ό,τι αφορά τι πιστώσει. Το ελεκτικό συνέδριο είπε ότι οι πιστώσει είναι νομικέ και κανονικέ σε όλε τι ουσιαστικέ πτυχέ. Πρόβλημα έχουμε σε επίπεδο πληρωμών. Εκεί στην τελευταία διαδικασία απαλλαγή είδαμε ότι το, ρυθμός λάθος, το ποσοστό λάθο είναι 3,9% και το DAS ε, ξεπερνά το επίπεδο σημαντικότητας. Τώρα θέλω να επικεντρωθώ στους λόγους. Τι πήγε στραβά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αν πάρετε τη γεωργία, που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι των δαπανών, αν ακούσετε τα κρατη λένε ότι εμείς έχουμε το ιερό δισκοπότηρο. Ε, καταγράφονται ε, ποσοστά ε, λάθος που είναι κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας, κάτω από το 2%. Στον πυλώνα 1, 0,55% ποσοστό λάθος. Για τον πυλώνα 2 μας λένε ότι το ποσοστό λάθος είναι 1,89%. Αλήθεια είναι αυτό. Η Κομισιόν έκανε τη δική της αξιολόγηση και κατέληξε επί τη βάση των εργασιών που έκανα αλλά και επί τη βάση των ε, ελέγχων του ελεκτικού συνεδρίου ότι δεν είναι αξιόπιστα αυτά τα δεδομένα. Υπάρχουν πάρα πολλά, προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλές αδυναμίες. Αυτό που έκανε η Κομισιόν είναι να θέσει έναν, ένα ανώτατο όριο 25%. Έχουμε δηλαδή 25% στο, προσέθεσε ένα 25% στο ποσοστό λάθο που είχε καταγραφεί για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Οπότε το 0,55% ε, των κρατών μελών γίνεται 0,69% για τον πρώτο πυλώνα και ε, από το 1,89% του δεύτερου πυλώνα των κρατών μελών πάμε πάνω από το όριο σημαντικότητα, πάμε στο 2,36%. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία με τα στοιχεία του ελεγκτικού συνεδρίου τώρα. Το ελεγκτικό συνεδρίο λέει ότι ο πρώτο πυλώνα ε, έχει ποσοστό λάθο 2,90%. Δεύτερο πυλώνα είμαστε στο 7,70%. Τώρα, η Κομισιόν πρέπει να δεχτεί και θα δείτε ότι έχει υπάρξει βελτίωση σε σχέση με το θέμα αυτό σε σχέση και με τις, τις εκθέσεις ε, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας για το 2012, ότι η γενική συνολική αξιολόγηση αυτού του τομέα πολιτικής δεν είναι επαρκής. Πρέπει να ξέρουμε πολύ, περισσότερα, λεπτο, πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σε επίπεδο διαφόρων αρχών πληρωμών, ε, αρχών πιστοποιήσεων ε, κτλ. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο για την γεωργία το οποίο εμπνέεται από τι ε, ε, γενικέ διευθύνσει που με τη συνοχή. Και θα σα εξηγήσω τι ακριβώ γίνεται εκεί. Θα ξεκινήσω με το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο τη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη, η οποία έχει στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά στοιχεία από τα εισαλλεκτικέ αρχέ των κρατών μελών. Μα παρουσιάστηκαν λοιπόν τα ε, συγκεκριμένα στοιχεία. 200, από 256 αρχές ε, μας είπαν ότι ο, ποσοστό λάθος είναι κάτω από 2%, για 69 υπηρεσίες 2 με 5% και μόνο για 15 το ποσοστό λάθος ξεπερνά το 5%. Αν το μεταφράσετε αυτό σε ένα χοντρικό υπολογισμό θα δείτε ότι δεν ξεπερνούμε το ε, όριο σημαντικότητας. Τώρα, η, τι έκανε η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ανέλησε ένα πρόγραμμα όλες τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της και κατέληξε στο εξής αποτέλεσμα. 35 ποσοστά λάθος είναι μη αξιόπιστα και 64 ποσοστά λάθος έπρεπε να επαναυπολογιστούν. Στο τέλος λοιπόν 69 επιχειρησιακά προγράμματα επηρεάστηκαν από πολύ υψηλότερο αριθμό λάθους, ποσοστό λάθους σε σχέση με αυτό που είχαν ανακοινώσει τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, για 25 τέτοια προγράμματα το ποσοστό λάθους ε, ήταν 10% και για 10 ε, προγράμματα το ποσοστό λάθους ήταν 25% ε, πάνω κάτω χρησιμοποιώντας την, τις καταποκοπή διορθώσεις. Συνολικά λοιπόν, ε, οι υπολογισμοί της ε, Κομισιόν δείχνουν ότι η δημοσιονομική, ο δημοσιονομικός αντίκτυπος ε, του προγράμμα του ποσοστού λάθους βρίσκεται στο 3, ανάμεσα στο 3,1 και στο 6,8 και αυτό είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που υπολόγισε το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο είχε πει ότι το ποσοστό λάθους βρίσκεται ανάμεσα σε 3 και 9% και κατά πάσα πιθανότητα το ποσοστό λάθους είναι γύρω στο 6%. Τώρα, Πάμε γρήγορα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Και μάλιστα επένασαν και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Μίλησαν για την κοινή προσέγγιση και από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από τα 117 ε, ποσοστά λάθους που ε, καταγράψαν τα κράτη-μέλη, μόνο 75 ε, έγιναν δεκτά, 20 προσαρμόστηκαν και 22 θεωρήθηκαν αναξιόπιστα ή μη καταγεγραμμένα. Στο τέλος λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τι πάει στραβά. Για να μην μακρηγορώ δεν λειτουργούν οι ενιαίοι έλεγχοι. Γιατί δεν λειτουργούν. Όχι γιατί δεν υπάρχει ιστορικό πλαίσιο ελέγχου που δεν ε, παρέχει διαφανή αποτελέσματα. Όχι. Δεν πάει καλά γιατί ένας ελεγκτής ε, δεν μπορεί να βασιστεί στον άλλο ελεγκτή. Δηλαδή τα κράτη-μέλη ε, διαβιβάζουν τα αποτελέσματά του, τα οποία όμω η Κομισιόν δεν μπορεί να δεχτεί, δεν μπορεί να τα δεχτεί ούτε το ελεγκτικό συνέδριο, οπότε κάτι δεν πάει καλά. Και δεύτερον, το, υπάρχει και το βασικό ερώτημα για το DAS. Η, τα, ελεκτικά, τα συστήματα ελέγχου και υποπτία είναι μερικώ αποτελεσματικά. Αυτό το έχει πει και το ελεγκτικό συνέδριο και βασίζεται στο δίκτυ ποσοστού λάθου. Έχει υπάρξει μια συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση για το αν έχει λόγο ύπαρξη η θετική δήλωση αξιοπιστία, η οποία όμω προβλέπεται από τη συνθήκη. Και σύμφωνα με τη συνθήκη, το δικαστήριο ε, πρέπει να παρουσιάσει μια γνωμοδότηση, το ελεκτικό συνέδριο πρέπει να παρουσιάσει μια ε, έκθεση συγγνώμη, για το αν ε, είναι νόμιμα και κανονικά τα στοιχεία. Και μάλλον αυτό είναι το λάθος που αποτρέπει την έκδοση της θετικής δήλωσης αξιοπιστίας. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν. Τα ελεκτικά συστήματα και τα συστήματα εποπτείας πρέπει να ενισχυθούν. 90% όλων των λαθών καταγράφονται εκτός κομισιών. Δηλαδή βρίσκονται σε επίπεδο τελικού αποδέκτη. Ο Μπράιον του είπε σαφέστατα ότι το, οι επίπεδοι πρώτου ελέγχου των κρατών μελών είναι αυτή που πρέπει να καταγράψουν και να διορθώσουν τα λάθη το ελεκτικό συνέδριο μας λέει και το επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα της Κομισιόν ότι για το ERDF 62 από τα λάθη που καταγράφηκαν από το ελεκτικό συνέδριο θα μπορούσαν να είχαν εξευρεθεί και από τα κράτη-μέλη στο κοινωνικό ταμείο 76%. Επίσης, άλλο ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την, α, τους αξιόπιστους δείκτες και, τα, αξιόπιστα στατιστικά, ε, στατιστικά στοιχεία. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ και για τον ενιαίο έλεγχο και είναι και προϋπόθεση για να βελτιωθεί το, το σύστημα. Αν η διάγνωση είναι λαθασμένη, τότε δεν υπάρχει, αν, δεν υπάρξει, ε, αν αυτό δεν αποτελεί λόγο αλλαγής του συστήματος, τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο τέλος. Επίσης, απλοποίηση. Ξέρετε ότι η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει μια ατζέντα απλοποίησης το 2012 για την ε, μετά την ε, εποχή, για, την εποχή μετά το 2013 και οι σχετικές διαπραγματεύσεις ε, που τρέχουν ακόμα επικεντρώνονται στη μείωση των αριθμών των προγραμμάτων, στην αναλογικότητα και στους ελέγχους σε σχέση με το κόστος να είναι αποτελεσματική και στην απλοποίηση των κανόνων επιλεξιμότητας και των μεθόδων κοστολόγησης. Η Κομισιόν έχει δημοσιοποιήσει τα scoreboards για την απλοποίηση και έχει αξιολογήσει την πρόοδο που έγινε. Κατά την άποψή μου τα αποτελέσματα σε κάποιους τομείς είναι ανησυχητικά. Θα μπορούσαμε να μην έχουμε καταλήξει σε ένα ενιαίο πλαίσιο, αλλά σε, ένα ίσως πιο περίπλοκο πλαίσιο. Τώρα, δύο λόγια για τους μηχανισμούς του διορθωτικούς ή προληπτικούς. Αναφέρθηκαν κάποια τελικά στοιχεία, θα ήθελα εγώ να σας πω. Αν δείτε τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις ανακτήσεις και τα προσθέσετε, καταλήγετε σε αριθμητικά στοιχεία ε, δείτε το μάλιστα και με τις συνολικές πληρωμές, ανάμεσα στο 1,7 και 1,4%. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε αυτό το κομμάτι από, τον από το ποσοστό λάθους που έχει προβλέψει το ελεκτικό συνέδριο, γιατί αυτές οι προβλέψεις διορθώνουν λάθη ε, από τα έτη νήμιον 1, νήμιον 2, νήμιον 3. Λαμβάνονται στο, στο έτος νη, αλλά αναφέρονται προφανώς σε, έχουν αναδρομική ισχύ. Ε, και τα, οι, οι, οι, ε, οι μελλοντικές που θα γίνουν θα γίνουν ε, για τα επόμενα χρόνια. Το, ε, αυτό που έχει προβλέψει το ελεκτικό συνέδριο είναι χρήσιμο και πρέπει να μπει στο μελλοντικό πλαίσιο. Και βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη από την Κομισιόν. Τώρα, τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Νομίζω ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός και το σχετικό άρθρο 32 είναι πολύ σημαντικά. Εάν το επίπεδο λάθο είναι ιδιαίτερο υψηλό, η Κομισιόν πρέπει να καταγράψει τις αδυναμίες στους, στα συστήματα ελέγχου, να αναλύσει το κόστος και το όφελος κάποιων διορθωτικών ε, μέτρων. Και επίσης, επί τη βάση αυτής της ανάλυσης, θα πρέπει να αναλάβει ή να προτείνει τις απαραίτητες δράσεις, δηλαδή απλούστευση, βελτίωση των συστημάτων ελέγχου, ή ανασχεδιασμό του προγράμματος ή του συστήματος παραδοτέων. Ξέρω ότι έχω ξεπεράσει λίγο το χρόνο μου, αλλά πρέπει να σας δώσω την απάντηση στο ερώτημα αν είναι ρεαλιστικό να έχουμε τελικά μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Κάτω από κάποιες προποθέσεις, ναι. Αν οι, τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας βελτιωθούν και γίνουν αποτελεσματικά, εάν οι δείκτες είναι αξιόπιστοι και επιτρέψουν σε όλους που πρέπει να δράσουν να δράσουν, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση, εάν υπάρξει απλούστευση, και εάν η, ο αντίκτυπος των προσπαθειών της Κομισιόν να προστατεύσει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ληφθούν υπόψη, τότε μπορεί να έχουμε το ιερό δισκοπότηρο στα χέρια μας στο εγγύς μέλλον. Εάν μία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρείται, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά, και αναφέρομαι εδώ σε αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, γιατί το 2% είναι πάρα πολύ δύσκολος στόχος να επιτευχθεί. Ειδικά λοιπόν, εάν κάποιο λάβει υπόψη του και τι ε, πολιτικέ λιτότητα και τη μείωση του προσωπικού, καθώ επίση και την αποτυχία τη εισαγωγή τη ε, απλούστευση για κάποιου τομεί. Αυτά από μένα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και λυπούμε που ε, δαπάνησα τόσο χρόνο. Yeah, thank you Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Ήταν δύσκολο να σα διακόψω γιατί εσείς ηγείστε στην Κομισιόν των υπηρεσιών που θέλουν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία προσδοκούμε από εσά. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε το ιερό δισκοπότηρο. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια του ουρανού βέβαια για να πετύχουμε το θετικό DAS. Θέλουμε βέβαια τη βοήθεια του ελεκτικού συνεδρίου και η κυρία Κάλιου Λάιντ ίσως μπορεί να μας βοηθήσει στο θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω το έργο των ελεκτών μπορεί να διευκολυνθεί και να απλοποιηθεί με αυτή την ε, πιο διάφανη διαδικασία που προτείνει ο κύριος Κράφτ. Θα ήθελα τώρα, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, να υπενθυμίσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Κομισιόν ζήτησε να υπάρξει αυτό το ελεκτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να βασίζεται σε ένα ενιαίο λογιστικό έλεγχο. Το 1994 η διαχείριση των ε, δημοσιονομικών των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινή διαχείριση έδειχναν μεγάλες αποκλήσεις. Η έλεγχη δεν ήταν παραπάνω, κάτι παραπάνω από μια αλληλεπίδραση ad hoc μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και κρατών μελών. Το σύστημα αυτό δεν είχε ιεραρχική δομή και δεν υπήρχαν αρκετοί έλεγχοι από τα κράτη-μέλη. Ήταν κυρίως η Κομισιόν και το Ελεκτικό Δικαστήριο ε, που ελέγχαν εκ των υστέρων αυτά τα οποία έκαναν τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό αφορούσε μονάχα ένα μικρό τμήμα των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ήταν κάτι που ίσχυε σε όλους τους τομείς. Η μεταρρύθμιση βέβαια στη Γεωργία οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις στις, στους ελέγχους των κρατών μελών. Το πρόβλημα ότι η Κομισιόν δεν ενσωμάτωσε τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων στην ανάλυση των τεκτενομένων. Ούτε η Κομισιόν άντλησε συμπεράσματα από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Συγχρόνως, όλη τη διαδικασία της δεκαετίας του 1990, ο λογιστικός και δημοσιονομικός έλεγχος έγινε σημαντικό εργαλείο <clears throat> για να αντιμετωπιστούν δημόσιες δαπάνε, να αυξηθεί η διαφάνεια και να διαχειριστούμε σωστά του κινδύνου. Σιγά σιγά αυτό οδήγησε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο εσωτερικών, εσωτερικού ελέγχου που με ένα πυραμιδικό τρόπο βασίζεται κάθε επίπεδο ελέγχου στο προηγούμενο. Και τα, σημεία, τα πρότυπα του Κόσο ήταν τα σημεία αναφοράς. Όλα αυτά τα πρότυπα έγιναν πολύ σημαντικά όταν ε, φτάσαμε στη δεκαετία του 2000, ιδίω σαν τμήμα της μεταρρύθμισης κοινοπτής Κομισιόν. Έτσι, η Κομισιόν οδήγησε σε ελάχιστε απαιτήσει από τα κράτη-μέλη για τον έλεγχο των διαφορετικών ταμείων. Ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να πιστοποιήσουν τι ε, αιτήσει επιστροφή από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τις, ε, τα ασθενή σημεία και του κινδύνου στο σύστημα. Να ελέγχουν τουλάχιστον 5% των δαπανών και να παρουσιάζουν μια δήλωση για κάθε πρόγραμμα το οποίο περατώνονταν. Δεν ήταν επαρκή όμω αυτέ οι αλλαγέ. Ετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία απαλλαγής του 2002, το Ελεκτικό Συνέδριο το 2004, στην γνωμοδότηση 2-2004, θέσπισε τις κύριες αρχές και τα κριτήρια για ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου μέσα στο κοινό πλαίσιο ελέγχου. Θεώρησε το Ελεκτικό Συνέδριο ότι υπάρχουν ορισμένε γενικέ αρχέ οι οποίε είναι κομβικέ για οποιοδήποτε εσωτερικό σύστημα ελέγχου το οποίο θέλει να καταλήξει σε ένα ενιαίο λογιστικό ε, έλεγχο μεθοδολογικά. Ποιε είναι οι γενικέ αυτέ αρχέ. Πρώτα απ' όλα, οι έλεγχοι θα πρέπει να βασίζονται σε κοινά πρότυπα και να είναι συντονισμένοι για να μην υπάρχει περιττή επικάλυψη. Αυτό είναι η αρχή της, του ενιαίου λογιστικού ελέγχου. Δεύτερον, οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται μέσα σε ένα ανοιχτό και διάφανο πλαίσιο με τρόπο που τα αποτελέσματά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα τμήματα του σύστηματος. Για μένα θα το έλεγα απλά ότι <clears throat> τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι διαθέσιμα σε όλους και αυτό είναι η έννοια της διαφάνειας στο λογιστικό έλεγχο. Ο στόχος λοιπόν κάποιου κάθε ενιαίου συστήματος θα πρέπει να είναι να είναι ενιαίο και να έχει το στοιχείο της διαφάνειας. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι πυλώνες του υποδείγματος αυτού. Το ελεκτικό συνέδριο επίση ανέφερε ορισμένου περαιτέρω πυλώνε που θα μπορούσαν να σταθεροποιήσουν αυτό το σύστημα. Η νομοθεσία πρέπει να είναι σαφή και απερίφραστη <clears throat> και να μην έχει περιττή πολυπλοκότητα. Επομένω να έχουμε σαφείς και καλώς καθορισμένους στόχους και προϋποθέσεις. Επίσης η Κομισιόν θα πρέπει να καθορίζει σαφή ελάχιστα πρότυπα και σαφείς στόχους για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τομέα όπου δαπανώνται κονδύλια. Αυτό θα βοηθούσε και το ελεκτικό συνέδριο να ελέγξει με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων το πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά. <clears throat> Επίσης, το ελεκτικό συνέδριο τόνισε και την, το αυξανόμενο κόστος των ελέγχων. Όταν η Κομισιόν σχεδιάζει σχέδια για δαπάνη να λαμβάνει υπόψη και το κόστος, τη σχέση κόστου κόστος-οφέλους για τα ελεκτικά συστήματα σε, διάφορα, σε τομείς του προϋπολογισμού. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτές τις ε, συστάσεις. Πρώτον, η νομοθεσία πρέπει να δίνει σαφείς και, κα... και απλούς στόχους. Δεύτερον, η Κομισιόν θα πρέπει να τις μεταμορφώνει αυτούς τους στόχους σε συγκεκριμένα ελάχιστα επίπεδα για τους εσωτερικούς ελέγχους. Και τέλος, όταν γίνεται ο σχεδιασμός των προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κόστος και η σχέση κόστος ωφέλειας των ελέγχων. Τόνισε επίση το ελεκτικό συνέδριο το να υπάρχει ένα υπόδειγμα ελέγχου, το οποίο να ευθυγραμμίζεται με τι αρχέ του ενιαίου ελέγχου, μπορεί να οδηγήσει στην μείωση των επικαλύψεων σε λογιστικέ έρευνε και να μειώσει και το διοικητικό άχθο για αυτού οι οποίοι είναι αντικείμενο λογιστικού ελέγχου. Ποια είναι τώρα η κατάσταση όμω τη εφαρμογή αυτών των κριτηρίων και των ωφελημάτων που μπορούμε να προσποριστούμε, όπω παραδείγματο χάρη μείωση του κόστου ελέγχου. Η πιο απλή απάντηση είναι βρισκόμαστε παρασάγκα μακριά από κάτι τέτοιο. Μπορώ όμω να το διαφοροποιήσω αυτό λιγάκι με το να σα παρουσιάσω ορισμένε πρόσφατε εξελίξει με τι αδυναμίε που είδε το συνέδριο στον τομέα τη πολιτική συνοχή. Όπου περνάει η διαχείριση από πολύπλοκου δέδλου. <clears throat> Στο χρονικό διάστημα 2013 το πλαίσιο ελέγχου είχε σαν στόχο ένα πιο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο με τρεις, τρία στρώματα εθνικού ελέγχου η αρχή διαχειριστική, η αρχή που πιστοποιεί και τελικά η αρχή λογιστικού ελέγχου. Η Κομισιόν είχε μεγαλύτερη ικανότητα να συμμετέχει στον έλεγχο αυτό με τη δυνατότητα να διακόπτει ή να αναστέλει πληρωμέ από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ύπαρξη ειδικών και ανεξαρτήτων λογιστικών αρχών ελέγχου ε, δημιουργήθηκαν και έπρεπε να παρουσιάσουν στην Κομισιόν ένα έλεγχο σε αντιπροσωπευτικό δημιουργηθηκαν και επρεπε να παρουσιασουν στην κομισιον ενα ελεγχο σε αντιπροσωπευτικο δειγμα προγραμμάτων, περίπου 400. Αυτό φυσικά αύξησε τον αριθμό των ελέγχων και το κόστος των ελέγχων, αλλά έτσι είχαμε το συμπέρασμα του, Συμβουλή, του Ελεκτικού Συνεδρίου τα τρία τελευταία χρόνια στις εκθέσεις του ότι έχει βελτιωθεί η διαχείριση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα συνοχής, παρά το γεγονός ότι το επίπεδο ατελειών είναι ακόμα ψηλό. Ο κύριος ε, λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα ελέγχου με την πλήρη δυναμικότητά του, όπω είπε και ο κύριο Κράφτη. Υπήρξαν πολλέ αστοχίε στα θέματα αυτά στα κατημέρια. Παραδείγματο χάρη, τα κατημέρια, που είναι η πρώτη γραμμή άμυνα εναντίον κατάχρηση <clears throat> των, ε, των δαπανωμένων κονδυλίων με έλεγχου στι αρχέ διαχείριση και πιστοποίηση. Το 2011, 60% τα σφάλματα που, των σφαλμάτων που εντόπισε το Συμβούλιο θα μπορούσαν να είχαν διορθωθεί και να εντοπιστεί από τα κράτη-μέλη. Είχαν επαρκείς πληροφορίες για τα θέματα αυτά. 2010 και 2011 βρήκε επίση το Ελεκτικό Συνέδριο ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να βασίζεται πλήρω και να εξασφαλίζεται από το έργο των Εθνικών Ελεκτικών Αρχών. Παραδείγματο χάρη, το πλαίσιο του ελέγχου δεν καλύπτει όλου του κινδύνου για ατασταλίε και ιδίω σε ό,τι αφορά τι δημόσιε προμήθειε και τι κρατικέ επιδοτήσει. Δεύτερον, η δειγματοληπτική μεθοδολογία δεν ακολουθούσε τι ε, κατευθυντήριε γραμμέ που είναι θεσπισμένε για τα θέματα αυτά και επίση δεν υπήρχαν στοιχεία σε σχέση με τα ασφάλματα προεκβολή και αξιολόγηση. Επομένω, υπάρχουν προβλήματα και ατέλειε που δεν αναφέρονται από τι εθνικέ αρχέ. Όλε αυτέ οι αδυναμίε μπορούν να είναι και αποτέλεσμα μιας εγγενούς ε, σύγκρουση συμφερόντων και εγγενών σφαλμάτων του κοινού συστήματος διαχείρισης. Για να είναι αποτελεσματικό αυτό το σύστημα και να παραμένει κάτω από το 2% θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να μπορέσουν να αποφευθούν οι δημοσιονομικές ε, διορθώσεις. Πολλές φορές οι αρχές τείνουν να υποτιμούν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται για να μην υπάρξουν αναστολές. Και αυτό έγινε πιο σαφές στην περίοδο 2000-2006. Οι έλεγχοι των πρώτων φάσεων της διαδικασίας περάτωσης των ελέγχων δείχνουν ότι για να μην υπάρξουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, οι αρχές των κρατών μελών παρουσιάζουν ποσοστά σφάλματος τα οποία ξεπερνούν τα τελικά ποσοστά ε, ε, σφάλματος χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως δικαιολογία. Τέλος, να δούμε τις επιπτώσεις για το κόστος. Οι ενισχυμένοι έλεγχοι του 2007-2013 έχουν αυξήσει σίγουρα αυξηθεί σίγουρα λόγω των αυξημένων ελέγχων. Θεωρούν ορισμένοι ότι το κόστος αυτό φτάνει το 0,2% του προϋπολογισμού συνοχής για το μέλλον. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα στοχευμένη δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν τα κράτη-μέλη αναλάβουν την ευθύνη και παίξουν σωστά το ρόλο του. Αλλά οι διαφορές στην εμβέλεια των ελέγχων και την έλλειψη, η έλλειψη ποιότητος ελέγχου δείχνουν ότι τα γενικά κριτήρια για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και έχουμε κάποιο δρόμο να διατρέξουμε. Θεωρώ τα άρθρα 31 με 33 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού είναι κινούμενα στη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι αυτά θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες απαιτήσει για το πλαίσιο 2014-2020, όπως εθνικές δηλώσεις διαχείρισης, πιστοποιημένες αιτήσεις εκθέσεις και γνωμοδοτήσει σε αιτήσει εκθέσει των ελεκτικών αρχών. Επίση, θα δώσει στην Κομισιόν δυνατότητα να έχει δεσμευτικέ κατευθυντήριε γραμμέ και να κάνει και δημοσιονομικέ διορθώσει. Από την άλλη πλευρά, η περισσότερη παραγωγή εκθέσεων δεν θα οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα δαπανών αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά τα στοιχεία αυτά από την Κομισιόν. Τα τελευταία δέκα χρόνια, δυστυχώ, η Κομισιόν έχει καταβιδιστεί κατά το βάρο των εκθέσεων των κρατών που πολλέ φορέ έχουν δημοσιευτεί χωρί την απαραίτητη επαλήθευση. Τέλος υπάρχει και μια εγγενή σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να υπονομεύσει το έργο της μετακύλησης του ελέγχου στις εθνικές αρχές αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα και το κατάλληλο σύστημα κυρώσεων. Μήπως είναι πιο μικρά τα θετικά στοιχεία της τροποποίησης του στοιχείου από την, τις κυρώσεις που μπορούν να προκύψουν αν κάποιος αν η Κομισιόν ανακαλύψει ότι δεν έχουν λειτουργήσει τα συστήματα αυτά των κλίντρων. Εάν λοιπόν το κόστος της γνώσης είναι πολύ ψηλό, υπάρχει το πάντα η δυνατότητα να δίνει κανείς λαθασμένα στοιχεία προς την Κομισιόν. Τελικά, το ερώτημα είναι θέλουμε να πάρουμε ε, εισιτήριο λεωφορείου που κοστίζει ένα ευρώ ή να ρισκάρουμε 100 ευρώ πρόστιμο εάν μας πιάσουν. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν και για το κόστος του ελέγχου. Ευτυχώς έχω και μια δεύτερη παρέμβαση σήμερα που θα προτείνω κάπως λιγότερο ζωφερές προτάσεις για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα το λόγο έχουν ε, οι βουλευτές για να κάνουν τις ερωτήσεις που θα ήθελαν. Ποιος θα θέλει να ξεκινήσει, η εισηγήτρια, κυρία Τσέσκοβα και μετά κύριο Γκάγερ. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη για να μπορεί να μιλήσει και ο συνάδελφος. Υποθέτω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι μπορούμε να ακούσουμε όλες αυτές τις απόψεις ε, γιατί ούτως ή άλλως ε, το θέμα αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια όλων των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της Κομισιόν ε, και σε ό,τι αφορά την έλεγχο των λογαριασμών και σε ό,τι αφορά την απαλλαγή. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για το μέλλον. Θα με ενδιαφέρει η άποψή σα σε σχέση με το εξή και τη Κομισιόν και του Ελεκτικού Συνεδρίου βεβαίω. Η Κομισιόν σκέφτεται να κάνει νέε προτάσει οι οποίε θα αντικαθιστούσαν αυτό το τρέχον σχέδιο δράση και ελπίζω ότι έχω καταλάβει καλά από την παρέμβαση του κυρίου Κραφ, του εκπροσώπου τη Κομισιόν, ότι θα επιτύχουμε μια αξιόπιστη δήλωση που μέχρι στιγμής ήταν ε, ανέφικτο να γίνει. Οπότε ερώτηματα προς το μέλλον. Ευχαριστώ. κύριος Γκάιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους πήραν το λόγο. Ήταν πραγματικά χρήσιμες οι παρεμβάσεις σας γιατί νομίζω ότι θέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύουμε και το περιγράφουν σαφώς, δείχνουν τι θα ήταν απαραίτητο να γίνει και σε ό,τι αφορά την ε, απαλλαγή, ώστε να βρούμε αυτό το ιερό δισκοπότερο που ψάχνουμε. Οι προοπτικές δεν είναι πολύ καλές, μάλλον θα πρέπει να γράψουμε την 19η, 20η, 21η έκθεση απαλλαγής μέχρι να έχουμε έστω και μία περιορισμένη αξιοπιστία, θετική δήλωση αξιοπιστία για την Κομισιόν. Βεβαίω αυτό θα έχει και πρακτικές συνέπειες για τη δουλειά της Επιτροπής. Ο κύριος Κράφ μίλησε για διάφορα γρανάζια που μπορούμε να κινήσουμε από κοινού με την Κομισιόν έτσι ώστε να προωθήσουμε αυτή την δήλωση αξιοπιστίας. Εγώ στη δική μου έκθεση απαλλαγή μίλησα πάρα πολύ για τι ε, ευθύνε των κρατών μελών. Βεβαίω υπάρχει και ευθύνη του Κοινοβουλίου. Η ευθύνη του Κοινοβουλίου, αγαπητέ Μάνφρεντ, το είπε αρκετά, το είπε ακροθυγό, ότι υπάρχουν κάποιε συμφωνίε, πλαίσια που δεν διευκολύνουν, ε, αλλά δυσκολεύουν την οικονομική διαχείριση. Αυτό βεβαίως ε, προκύπτει από, από το Κοινοβούλιο, γιατί και εμείς έχουμε ε, την ευθύνη μας. Αν περιπλέκονται τα ταμεία, τότε προφανώς και ο έλεγχος των ταμείων θα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο και προφανώς και τα λάθη θα είναι πολύ περισσότερα. Γι' αυτό το ερώτημά μου έχει να κάνει με το scoreboard. Είναι δυνατόν η Κομισιόν στο σύνολο του να, να ενημερώνει το σύνολο του Κοινοβουλίου για το τι γίνεται με τα scoreboards στην Κομισιόν. Πότε αυτά ξεπερνώνται και πότε όχι. Γιατί το ελάχιστο που θέλουμε εμείς είναι οι επιτροπές που ακριβώς δουλεύουν πάνω σε αυτά τα πλαίσια να γνωρίζουν αν κάνουν ένα σωστό πολιτικό βήμα προς τα εμπρός ή αν απλώς περιπλέκουν τους ε, κανόνες ε, που τελικά θα μας οδηγήσει σε περισσότερα, ε, σε περισσότερα λάθη. Οπότε το θέμα είναι η Κομισιόν ας μην κομίσει γλαυκές Αθήνας. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα κυλήσουν και οι διαπραγματεύσεις. Προφανώς θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια. Έχουμε μία ευκαιρία να επηρεάσουμε την ε, συμφωνία πλαίσιο. Έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κίνδυνο αύξηση των ποσοστών λαθών. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς, ε, ερωτήσεις υπάρχουν. Κατά πρώτον, είναι αδύνατον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εναρμονίσει τι πρακτικέ που ακολουθούν οι υπηρεσίε τη. Πραγματικά, αν υπήρχε πολιτική βούληση και αν ο πρόεδρο τη Επιτροπή πίεζε, ασκούσε πίεση, νομίζω περισσότερα θα πετυχαίναμε. Αυτό είναι μια πεποίθηση ειλικρινή δική μου. Και εάν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είστε πεπισμένοι ότι δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, δεν θα έπρεπε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή στα κατήμελη μια αλλαγή στη συνθήκη. Δεν θα ήταν αυτή μια διέξοδο, η αλλαγή τη συνθήκη. Και αντικατάσταση τη της ε, θετική δήλωση από μια προσέγγιση που να βασίζεται στη μέτρηση των επιδόσεων. Οπότε δεν θα επιφορτίζονται αποκλειστικά και μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, το βάρο του έργου. Καταλαβαίνω ότι ξεπερνά τι αρμοδιότητε του κ. Κράφ αλλά είμαστε σε δημόσια ακρόαση, οπότε μπορεί ο καθένα να πει την προσωπική του άποψη. Και κάντε κι εσεί το ίδιο, παρακαλώ. Thank you, Chairman. I will... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τη δική σας ερώτηση, η οποία είναι εκτενέστατη. Ξέρετε ότι ανά τον κόσμο δεν υπάρχουν πολλές συνταγματικές διευθετήσεις που να προβλέπουν κάτι τέτοιο σαν την ε, δήλωση εξοπιστίας, τον ΤΑΣ. Είμαστε μια εξαίρεση σε αυτό. Και νομίζω ήδη ακούστηκαν στο παρελθόν σχόλια της σκέψης για το ότι θα έπρεπε να αλλάξει η συνθήκη. Όμως, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολιτικές συζητήσεις, όπως έχει ήδη συμβεί με το ΝΤΑΣ, διότι λένε τώρα δεν μπορούν να, να κάνουν αυτά που υποσχέθηκαν, οπότε πάλι αλλάζουν ε, το τέρμα. Δεν μπορούν να βάλουν γκολ και αλλάζουν τη θέση. Εγώ είμαι λιγότερο πολιτικός και περισσότερο ε, τεχνικός εμπειρογνώμων, για να το πω έτσι. Ήταν πολιτικό το ερώτημά σα. Εγώ νομίζω οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα χαίρονταν μάλλον οι Ευρωπαίοι πολίτε θα χαίρονταν αν εξαφανιζόταν από τη συνθήκη των ΤΑΣ. Διότι ένα από του προηγούμενου ομιλητέ ρώτησε τι είναι πιο σημαντικό, η περισσότερη συμμόρφωση ή οι καλύτερε επιδόσει. Για μένα προφανώ είναι οι καλύτερε επιδόσει η απάντηση. Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι κανόνε συμμόρφωση και αιρεσιμότητα πρέπει να διασυνδέονται με τι επιδόσει. Αλλά βεβαίω μόνο σε ένα τέλειο κόσμο. Ξέρουμε όμω ότι στην πράξη αυτό συνήθω δεν συμβαίνει. Και επίση τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια συνεπέστερη προσέγγιση μεταξύ των υπηρεσιών τη Επιτροπή. Εδώ να πω ότι υπήρχαν διαφορετικές κίνδυνοι και πιέσει ε, στι υπηρεσίε τη της Κομισιόν, αποκεντρωμένη διαχείριση, ε, κοινή διαχείριση, κοινή διαχείριση του κινδύνου και ούτω καθεξής. Ε, η λύση η ενιαία για όλους θα ήταν κάτι το δύσκολο να εφαρμοστεί. Υπάρχει ένα λοιπόν κοινό πλαίσιο με κοινά στοιχεία που θα μπορούσε να εξυπηρετεί τους πάντες, αλλά υπάρχουν, υπάρχει δυσκολία των λεπτομεριών που είναι δαιμονικές καμιά φορά. Θα έπρεπε λοιπόν να προσαρμόσει κάποιο κάποια στοιχεία στους διαφορού τομεί αναλόγω με το τι χρειάζονται. Για το πολύ σημαντικό ερώτημα της απλούστευση, τον ε, πίνακα αξιολόγηση. Οι δύο πίνακε που έχει οθετήσει ω τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτού του τύπου είναι δημόσια έγγραφα και δίνουν διαφανέστατε πληροφορίε για το ποια ήταν η αρχική πρόταση, ποιο ο επιδιωκόμενο στόχο και πού έχουμε φτάσει στην όλη συζήτηση. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι απλώς δημοσιοποιεί και το τι επιδιωκόταν και το τι κίνδυνοι υπάρχουν, ε, εκτός βέβαια αν δεν υπάρχουν αρκετά καλοί δείκτες ή υψηλότερα ποσοστά στο μέλλον. Για τη δική σας ερώτηση, κυρία Τσέσκοβα, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει άλλο πρόγραμμα δράσης από προσωπική άποψη, γιατί δεν έχει συζητηθεί ακόμη στο επίπεδο του δικού μου φορέα, για μένα το άρθρο 32, εδάφιο 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, είναι το ιδανικό μέσο. Εάν δούμε ότι έχουμε ψηλό ποσοστό σφαλμάτων και το βλέπουμε σε πολλούς τομείς πολιτικής, τότε πρέπει να διερωτηθούμε τι πρέπει να γίνει για να ε, βελτιωθεί η κατάσταση, να μετρήσουμε το κόστος των μέτρων που θα προτεθούν και το όφελος που μπορεί να προσφέρουν. Νομίζω ότι στην όλη συζήτηση και με τους εκπροσώπους της Επιτροπής σας και του σώματος σας του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και με το Συμβούλιο θα μπορούσαμε να επιτελέσουμε πρόοδο ώστε να βελτιωθεί ε, παρκώς η κατάσταση. Και πάλι να υπογραμμίσω. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι το όριο της Το όριο της σημαντικότητας είναι 2%. Επίσης και η έλεγχη των, ε, της αποτελεσματικότητας είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και η ανάγκη να, προστατευτεί, να, να προστατευτούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Έτσι θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο είπε ο κύριο Γκάιερ είναι πολύ σωστό. Ε, με αυτό που είπα για την διαχείριση βάση ισοών και τόνισε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα περισσότερη από το προηγούμενο σύστημα. Θα είναι ένα ευρυντικό σύστημα που να βασίζεται και σε εισρωές και σε εκροές στο, στη διαχείριση. Βρίσκομαι τώρα στα χέρια των νομοθετών για τα θέματα του ελέγχου και η επόμενη παρουσίασή μου είναι πώς να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια καλύτερη απόδοση στα θέματα αυτά. Άκουσα ότι ο κύριος Κράφτ πιστεύει ότι ίσως το ίδιο το DAS, θα, το πιστοποιητικό αξιοπιστίας, δεν θα πρέπει να υπάρχει στις μεταρρυθμισμένες συνθήκες. Εδώ έχω μια κάπως διαφορετική άποψη. Νομίζω το κύριο πρόβλημα με το πιστοποιητικό αξιοπιστίας από την αρχή είναι ότι ζητούσε μονάχα από το ελεκτικό συνέδριο να δώσει αυτό το πιστοπικό αξιοπιστίας, αλλά όχι ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου να ξεκινά από τα κράτη-μέλη μέχρι το ελεκτικό συνέδριο. Οπότε δεν υπάρχει η αλυσίδα αξιοπιστίας. Ε, αυτή, ε, δεν υπήρχε καταρχήν η αλυσίδα αξιοπιστίας, η οποία τώρα δημιουργείται σιγά-σιγά και έρχεται στη ζωή. Πιστεύουμε ότι το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στο τι κάνουν τα κατημέρια και το τι κάνει η Κομισιόν. Με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσουμε τους πόρους που χρησιμοποιούμε και θα μπορέσουμε να φέρουμε το υπόδειγμα του ενιαίου ελέγχου στην πραγματικότητα. Δυστυχώς γεννήθηκε επταμινήτικο το ΝΤΑΣ και η ιστορία επαναλαμβάνεται και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η συζήτηση για την ad hoc εκτίμηση της απόδοσης. Θα όμως στην επόμενη παρέμβαση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Θα έλεγα να συνεχίσουμε όμως τώρα με την ακρόασή μας και τώρα θα καλέσω τον Ζουλ Μουίς να έρθει εδώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κράφτ. Έχουμε εδώ πέρα την ανάγκη να αλλάζουμε καρέκλες, είναι ένα παιχνίδι με μουσικές καρέκλες επειδή είναι λίγες οι θέσεις στα προεδρικά έδρα και πρέπει να αλλάζουν θέση οι εμπειρογνώμονες. Κύριε Μούης, χαιρετώ, σας χαιρετώ, χαιρετώ την έλευσή σας και είστε στο παρελθόν επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναφερθείτε στο θέμα του αν το πιστοποιητικό αξιοπιστίας είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ένας πραγματικός έλεγχος και ποιες είναι οι δυνατότητες μιας πιο αποτελεσματικής ε, ε, αξιοπιστίας που θα εμπλέκει και τους πολίτες. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, οι προηγούμενοι ομιλητέ και ιδίως η συγκεκριτή κυρία Τσέσκοβα διευκόλυναν πάρα πολύ το έργο μου. Έγιναν ήδη σημαντικές παρατηρήσεις σήμερα Ιδιαίτερος διότι όλοι φαίνονται να κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Μία είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ μου και των υπολείπων ομιλητών. Οι περισσότεροι επιχειρηματολογούσαν υπέρ της ε, εξέλιξης. Εγώ θα προτιμούσα την επανάσταση για να το πω έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο κλειδί και θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε ένα σωστό πλαίσιο ευθύ εξ αρχής γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ώστε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, ε, στο σημείο εισόδου εννοούμε τι ευθύνε των ε, κρατών μελών με, τις, ε, με τα δικά του πιστοποιητικά και τι δικέ του δηλώσει, ενώ το αποτέλεσμα είναι ο εξωτερικό έλεγχο και το πώ έχουμε εθιστεί σε αυτό που ονομάζουμε πιστοποιητικό αξιοπιστία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διαλύσω ένα μύθο, ο οποίος επανειλημμένος επανέρχεται εδώ οι ιδρυτές της ΕΚΑΧ ποτέ, μα ποτέ, δεν ζήτησαν ούτε επιδίωξαν το πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Ζήτησαν ένα πιστοποιητικό, αλλά όχι αυτό. Το πρόβλημα με τα λογιστικά και τον λογιστικό έλεγχο είναι ότι μόλις αποκτήσει κανείς ένα σύνολο κανόνων, αυτό γίνεται γλώσσα και μετά γίνεται και μια πραγματική κουλτούρα. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς τους ανθρώπους από τις συνήθειές του, γιατί υπάρχουν ε, βασικές συνήθειες και κοινά συμφέροντα. Όμως δεν νομίζω ότι οι συντάκτες της, ε, των συνθήκων, οι ιδρυτές του ελεγκτικού συνεδρίου, αν βλέπαν τη σημερινή κατάσταση και πόσο περίπλοκα έχουν γίνει τα πράγματα, πώ έχουν εξελιχθεί και αλλάξει, πόσες δυνατότητες υπάρχουν, ότι τα κράτη-μέλη πολλές φορές φεύγουν των ευθυνών τους. Θα χόρευαν στους τάφους τους. Αυτό που λένε λοιπόν εδώ οι ομιλητές είναι αυτό που ζητάμε κι εμείς σε ένα βαθμό, είναι να δοθεί έμφαση από κοινού από τα κράτη-μέλη στο θέμα των ευθυνών που τα ίδια έχουν. Αυτό που, θα που προσπάθησα να κάνω με το κείμενό μου είναι και πάλι να δώσω έμφαση σε κάτι που λέγεται τα τελευταία 7-8 ε, χρόνια και επαναλαμβάνεται ετησίως. Έχει γίνει κάτι που μοιάζει με ένα όνειρο που βλέπει κανείς ξανά και ξανά. Μια εμπειρία ήδη που την έχει φανταστεί. Μια ψευδέστηση διότι πρέπει να παρακολουθούμε και τις πολιτικές εξελίξεις. Αλλά τίποτε δεν θα έπρεπε να εμποδίσει την μετατόπιση του συστήματος που χρησιμοποιούμε και τη βελτίωσή του. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ σε δύο στοιχεία. Την βελτίωση στο επίπεδο της ε, αρχής της διαδικασίας και του τέλους τους. Έχω αφήσει βέβαια κατά μέρο τη μέση, διότι θα ήθελα να είχα συμμετάσχει στο προηγούμενο πάνελ, ε, στην προηγούμενη συζήτηση για τη δημοσιονομική στήριξη. Στην Παγκόσμια Τράπεζα, όπου εδώ και πέντε χρόνια εργάζομαι ως ελεγκτή, διαφορά, συζητήσαμε την ε, διαφορά μεταξύ εκθέσεων προγραμμάτων και εκθέσεων ε, προπολογισμού. Υπάρχουν δύο παράλληλε οδοί εδώ και κάτι που θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε για τη δική μας δημοσιονομική στήριξη από τη σκοπιά των προγραμμάτων και το πόσο αυτά διαρθρώνονται και οργανώνονται και πώς διαδικαστικά ε, καταρτίζονται για το Ταμείο Συνοχής λόγου χάρη για τα γεωργικά ταμεία. Τα έχω πει και στο παρελθόν. Έχω ταχθεί υπέρ του να μην τα ονομάζουμε καν στήριξη προγραμμάτων, αλλά δημοσιονομική στήριξη. Αν θέλουμε να έχουμε, αν θέλουμε μάλλον να έχουμε τη δυνατότητα να μετατοπίζουμε κονδύλια μεταξύ των χωρών και έχουμε τόσο μικρό περιθώριο πολιτικών ελιγμών, μιλάμε πλέον για δημοσιονομική στήριξη και όχι για κάτι άλλο. Για, για τα εθνικά πιστοποιητικά. Είχα αναφέρει και προτείνει, αν δεν το πιστεύετε, ήδη από το 2001, στην πρώτη συνάντηση εσωτερικών ε, λογιστών ελεγκτών, Είχα κάνει δύο προτάσει και το 2005 το Κοινοβούλιο νομίζω τι υιοθέτησε. Αν οι βασικοί φορεί ήταν οι εθνικέ κυβερνήσει και αν οι εθνικέ κυβερνήσει ήταν και ε, ο πιστωτή και ο, ο φιλέτης, τι άλλο, τι πιο λογικό από το να ζητά κανεί να λογοδοτήσει. Να λογοδοτήσουν οι ίδιοι. Και τα πάντα να καταγράφονται σε εκθέσει όπω δει. Ήταν ε, μια περίοδος αρκετά ταραγμένη από τότε. Τρεις-τέσσερις χώρες μόνο προσφέρθηκαν ε, να το εφαρμόσουν αυτό και από αυτές τις τέσσερις χώρες εξ όσων γνωρίζω, καμία, καμία δεν, την, δεν ε, φρόντισε την ακρίβεια για και την πληρότητα ως προς τη συνεισφορά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως Ευρωπαίος πολίτης, ως φορολογούμενος. Και για κάποιον που έχει περισσότερο χρόνο να διαβάζει εφημερίδες ή blog στο ίντερνετ και ούτω καθεξής. Φανταστείτε να σκέφτεται οποιαδήποτε χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται βοήθεια και να πηγαίνει να λέει στην κυβέρνηση ζητάς από τους πολίτες σου να ε, από τις δικές τους φορολογικές επιστροφές να ε, αφιερώσουν κάποιο ποσό τις φορολογικές τους απαλλαγές θες να τις ε, εγκρίνουν οι ίδιοι, οι ίδιοι να πιστοποιούν ότι είναι πλήρης φορολογική τους δήλωση. Τι τους κάνεις. Κάπως έτσι έχει γίνει και η κατάσταση με τις εθνικές ε, δηλώσεις και τα εθνικά πιστοποιητικά. Οι εθνικές κυβερνήσεις αρνούνται να ε, λογοδοτήσουν για το πιο την πιο θεμελιώδη αρχή που θα έπρεπε να ισχύει από την πλευρά της λογοδοσίας για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη δική τους τη συνεισφορά προς αυτήν. Δεν ξέρω πώς το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μπορεί να εγκρίνει την πληρότητα των εισοδημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν οι βασικοί πρωταγωνιστές δεν θέλουν, δεν μπορούν ή δεν πρόκειται να ε, λογοτήσουν και τα εισοδήματα. Δεν βλέπω λοιπόν καμιά άλλη επιλογή, και εδώ ερχόμαστε στην έννοια τη επανάσταση, καμιά άλλη επιλογή ε, πέραν των εθνικών πιστοποιητικών. Εάν δεν μα στείλει εθνική δήλωση του χρόνου, δεν θα σου στείλουμε χρήμα. 10% έκπτωση, 20% μείωση, αλλά ο μόνο τρόπο να υπάρξει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στο σύστημα είναι αυτό. Και έτσι φτάνουμε στο τελικό σημείο, στο τέλος της διαδικασίας, την εξωτερικό, τον εξωτερικό έλεγχο, την, το πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Εν τω μεταξύ, παρεμβάλλεται ένα τεράστιο ποσό καλού έργο και εδώ χαιρετίζω τον ε, συνεργάτη μου, ο οποίος μαζί με τη στήριξη του Κοινοβουλίου και της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβάλλει σε όλα αυτά, τον κύριο Γκρέι, αλλά τα καλά νέα είναι ότι κανένας, ούτε οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκή Ένωσης, ούτε οι συντάκτες των συνθήκων, κανείς δεν ζήτησε το πιστοποιητικό εξοπιστίας όπως το ξέρουμε σήμερα. Είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε ελεύθερα, διότι το πιστοποιητικό αυτό έχει προσφέρει πολλά τα τελευταία 10-15 χρόνια, προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος και η σχετική ευαισθητοποίηση για τον έλεγχο. Αλλά πέρα από το ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να προσπογράψουν τέτοια έγγραφα, τίποτα δεν δικαιολογεί να έχουμε μια τέτοια διαδικασία που είναι τόσο γραφειοκρατική, ε, η οποία είναι από στατιστική άποψη πολύ λίγο αξιόπιστο από την εποχή της ΕΚΑ και δεν δικαιολογείται από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚ, οι οποίοι έχουν τέτοιο δημοσιονομικό σύστημα που λειτουργεί επαρκώς και ενώ ξέρουμε ότι έχουμε τέτοια σφάλματο, σφάλματος, 2,5-3,5 δεν με νοιάζει. Ίσως να μην το έχετε ακούσει σε προηγούμενες ομιλίες μου, αλλά απλώς έχω ιδιάσει με το πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Και νομίζω το ίδιο και εσείς θα έπρεπε να αισθάνεστε. Εάν πιστεύετε ότι σας προσφέρει κάτι καινούριο, πρέπει να σκεφτείτε πώς θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τον πιστοποιητικό αξιοπιστίας από το 2018. Πάλι θα συζητάμε για ποσοστίες μονάδες, ενώ αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε να βρούμε το ποσοστό των σφαλμάτων και είναι εκατοντάδες αυτοί που ψάχνουν τα ποσοστά. Καταργήστε το, καταργήστε το. Ήδη το λέει η συνθήκη. Η ΕΤΑΚ έχει την δυνατότητα το ελεγκτικό συνέδριο μάλλον έχει τη δυνατότητα να πάει σε εξωτερικούς ελέγχους και νομίζω ότι ενώ μιλάω κάποιο προσπαθεί να μου στείλει και κάποιο μήνυμα. Ε, στην όλη διαδικασία λοιπόν αυτή πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα από αυτά που απαιτούνται από το πιστοποιητικό αξιοπιστία, αλλά πουθενά η συνθήκη δεν λέει ότι πρέπει να εφαρμόζουμε το ε, πιστοποιητικό όπω το ξέρουμε. Και δεν ήθελα να κλείσω με αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μουής. Δεν ξέρω αν, αν βγαίνει στο ίντερνετ η παρέμβασή σας, ίσως κάποιος να ήθελε να σας δώσει τα άμεσα αποτελέσματα των όσων είπατε. Η κυρία Κάλγιουλαϊτ. Τα είπε ήδη ο κύριο Μή, ακούσατε τι σα είπε. Είπα και εγώ κάτι παρόμοιο στην ε, απάντηση που έδωσα στο προηγούμενο πάνελ. Οπότε πραγματικά συγχαίρω τον ε, κύριο Μουής και χαίρομαι που είμαστε και στο ίδιο μήκο κύματο. Όπω είπα στην προηγούμενη παρέμβασή μου, την τελευταία δεκαετία έχουν υπάρξει βελτιώσει στο σύστημα τη παροχή ε, κοινωνικών κονδυλίων. Το σύστημα αυτό έχει συγκεκριμένες ε, διαδικασίες για τους, ελεκτικούς, ε, για τους ελέγχους, αλλά όπως έχει πει το ελεκτικό συνέδριο, οι συνέπειες της διάπραξης λάθους είναι σημαντικές ε, γιατί δεν γίνονται οι εργασίες σύμφωνα με τα τρέχοντα κριτήρια γιατί υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων κριτηρίων. Οπότε το ερώτημα τίθεται για το κατά πόσο το τρέχον ε, ε, δύσκολο σύστημα στη διαχείρισή του μπορεί να δώσει ένα θετικό πιστοποιητικό αξιοπιστία συν το επιπλέον κόστος του, των επιπλέον ελέγχων. Στην ε, γνωμοδότηση 6-2010 για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, το, το ελεκτικό συνέδριο τόνισε ότι θα υπάρξουν, υπάρχουν κάποιε επιλογέ σε περίπτωση που είναι αδύνατο να υπάρξει υψηλό επίπεδο συμμόρφωση. Α πούμε, ε, απλούστευση των ε, κανόνων, ε, ανασχεδιασμό του προγράμματο, πιο στενή έλεγχη, ανοχή ενό υψηλού επίπεδου μη συμμόρφωση ή ε, πάυση τη δραστηριότητα. Η Κομισιόν έχει κάνει κάποιο πρόοδο στην απλούστευση των κανόνων και στην στους ελέγχους που κάνει, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι επαρκές. Υπάρχουν κάποια δείγματα που λένε ότι η Κομισιόν θέλει να αποφύγει το παρόν σύστημα και το ε, μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 παρέχει κάποιε δυνατότητε για να συνδεθούν οι πληρωμέ με τα αποτελέσματα. Τα κράτη-μέλη μπορούν από μόνα του να διαχειριστούν ένα, μια δέσμη προγραμμάτων σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ή κοινέ δράσεις, ε, κοινές, σχέδια Αυτό είναι ένα καλό βήμα, αλλά τα ε, κίνητρα είναι αντίθετα με το, το, σύστημα. Υπάρχει κίνδυνο η απόδοση να το σύστημα βάλων που βασίζεται στην απόδοση να, δώσει, ε, να συμπληρώσει απλώς ή να ε, αντικαταστήσει τις ε, παραδοσιακές μεθόδους. Επίση να πω ότι για τον τομέα τη έρευνα, η Κομισιόν έχει εισαγάγει τη δυνατότητα ε, χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστου ε, και ο το 2020 κάνει ένα βήμα παραπέρα για την ε, χρήση καταποκοπή ποσών για συνολικά προγράμματα σε συγκεκριμένου τομεί. Αν τώρα αυτή η πρόταση θα γίνει δεχτή από του δικαιούχου, θα το δούμε. Αλλά εμεί έχουμε ήδη κάποιε αμφιβολίε, αν δούμε και την εμπειρία που έχουμε κερδίσει με την χρήση των απλουστευμένων επιλογών λόγων για τα προγράμματα του ε, προγράμματος πλαισίου 7. Ο ελέφαντας παραμένει στο δωμάτιο. Τα κράτη-μέλη θα, παρα, θα πάρουν τον, ε, το ρίσκο να συμπληρώσουν τις ε, παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης με, χωρίς να αλλάξουν δραστικά την διαχείριση των εθνικών τους κονδυλίων. Θα πάρουν το ρίσκο να εφαρμόσουν ένα νέο συμπληρωματικό σύστημα εάν αυτό παραμείνει εθελοντικό. Υπάρχει κίνδυνος να χάσουν κονδύλια και υπάρχουν και κίνδυνος να γίνουν λάθη στα πλαίσια ε, του τρέχοντος συστήματος. Τώρα, ας δούμε τι είδος ε, αποτελέσματα ε, θα καταγράψει το ελεγκτικό συνέδριο στις, ε, στους ελέγχους συμμόρφωσης, όπως είναι το ΝΤΑΣ, σε περίπτωση που ισχύσει το ιδεατό, το ιδεατό σενάριο. Ένα πρόγραμμα διαχείρισης με βάση τα αποτελέσματα. Αν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει τη συμφων... την συμμόρφωση οδηγήσουν σε αποτελέσματα, θα οδηγηθούμε προφανώς σε μια αξιολόγηση επίδοσης και το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορεί να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για την επίδοση επίτευξη των στόχων της πολιτικής στα πλαίσια του, των ελέγχων του ΝΤΑΣ. Αν η, αν βεβαίω το πρόγραμμα βασίζεται στι επιδόσεις ή στην επίτευξη των στόχων. Για το 2012 και μετά, το ελεγκτικό συνέδριο δεν ελέγχει τι ε, πληρωμέ ε, πριν αυτέ αποδείξουν την οικονομική του ε, εφικτότητα. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει και τι δηλώσει μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους των ε, προγραμμάτων. Και αυτή η αλλαγή ήταν δυνατή μόνο επειδή η Κομισιόν έχει εφαρμόσει σε ε, παρκές επίπεδο την αλλαγή από, τις, από το σύστημα χρήσης μετρητών στις, στο σύστημα χρήσης των λογαριασμών. Μετά από αυτή την αλλαγή, το ελεγκτικό συνέδριο και η σχετική μεθοδολογία θα πρέπει να κρίνει ποιοι είναι οι, ε, οι στόχοι. Αν, ε, η, αν πληρείται η προπόθεση των πληρωμών, ε, τότε μπορούμε να το ελέγξουμε. Αν ε, το θέμα είναι η διαδικασία, μπορούμε και αυτό να το ελέγξουμε. Το θέμα ε, όμω είναι να δούμε κατά πόσο όλα αυτά συνάδουν και με τα όσα προβλέπει η συνθήκη. Στην, στο όραμα που έχουμε για τον 21ο αιώνα, για τους κανόνες και τους κανονισμούς, θα πρέπει να ε, αποφύγουμε περίπλοκους κανόνες γιατί κανένας δεν ε, μπορεί να ε, τους εφαρμόσει. Οι ελεγκτές βεβαίως πρέπει να παίξουν το παιχνίδι σύμφωνα με τους κανόνες. Η Κομισιόν λοιπόν είναι αυτή που θα προτείνει ένα καλύτερο πλαίσιο για, την, για τις ευρωπαϊκές δαπάνες και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσει πάνω σε αυτές τις προτάσεις. Πάμε τώρα ένα βήμα παραπίσω. Το τρέχον σύστημα βασίζεται σε συμβολή. Είναι ένα σύστημα όπου η προσοχή τίθεται στην ε, δημοσιονομική εκτέλεση και στα ε, ποσοστά απορρόφησης. Και για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε περαιτέρω, μάλλον πρέπει να επιβάλλουμε περαιτέρω απαιτήσει που θα σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων με, χωρίς να γίνει συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο μετά ανάμεσα στους ε, κύριους εμπλεκόμενους φορείς για το ποια είναι τα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε με την ε, ε, παροχή αγαθών και υπηρεσιών δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ε, προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα. Ήδη έχουμε μία προειδοποίηση για την μέτρηση της επίδοσης μόνο για χάρη της μέτρησης δεν είναι η Κομισιόν μόνο και δεν είναι δικό της το λάθος που το κείμενο περιλαμβάνει πάρα πολλές προφορίες για τις δαπάνες ε, που έχουν, ε, συγκεκριμένα, που έχουν πάρα πολλά δεδομένα ε, αμφιβόλου ποιότητας και σχετικότητας με το θέμα και δεν έχει και νόημα να πηγαίνουμε και να κάνουμε τη μέτρηση της επίδοσης χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα, συγκεκριμένους δείκτες. Θεωρητικά αυτά βεβαίως υπάρχουν, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται και τα αποτελέσματα δεν είναι ιδέατα. Ένα σαφή ορισμό του τι είδου πληροφορίε χρειάζεται το σύστημα είναι απαραίτητο. Να το να δημιουργήσουμε το πρώτο βήμα, να κάνουμε μάλλον το πρώτο βήμα, είναι προφανώ μια πρόκληση. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώ παίρνουν ω αντίκρισμα για τα ποσά για τα οποία φορολογούμε του Ευρωπαίου πολίτε. Οι δικαιούχοι όντω ωφελούνται από τα προγράμματα χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η θέση των ε, δικτών και των ε, στόχων θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε σχέση και με το τι γίνεται και ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη επίτευξη των στόχων. Το σύστημα πρέπει λοιπόν να είναι ευέλικτο για να μπορεί να περιλαμβάνει και τις διάφορες δυσκολίες που προκύπτουν. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τους στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας πούμε, το Connecting Europe ή κάτι παρόμοιο απόλυτα σαφές και αποδεκτό αξίζει τον κόπο να εφαρμοστεί μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Πρέπει όμως να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι στον προπολογισμό όπου αυτοί οι στόχοι δεν είναι απόλυτα προφανείς. Οπότε αυτοί οι τίτλοι του προπολογισμού δεν ακολουθούν την αρχή της επικουρικότητας και δεν θα πρέπει να βρίσκονται στον προπολογισμό αν τα επίπεδα στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι προφανή, είναι προφανώς αδύνατο να ε, υπάρξει κατανομή σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να ε, εκλογικεύσουμε τον τρέχοντο προπολογισμό. Με μια τέτοια σταδιακή προσέγγιση είναι, ε, είναι πιο εύκολο η Κομισιόν να καταλήξει σε μια προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό ακόμα απέχει πολύ. Δεν υπάρχει πανάκια για να λυθεί η πολιτική ε, συμφωνία για να περιορίσουμε πρώτα ε, τις ε, σφαίρες στις οποίες θα δουλέψουμε είναι αυτό που χρειάζεται. Χρειάζεται λοιπόν άλλα τέσσερα ή πέντε χρόνια να δημιουργήσουμε το σύστημα και μετά να το εποπτεύσουμε. Δεν είναι μόνο οι λεπτομέρειες που θα πάρουν χρόνο, αλλά είναι το θέμα της αλλαγής του πώς λειτουργούν οι διαχειριστές και πώς παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας. Και βεβαίως Όλα αυτά μπορούν να ξεκινήσουν ε, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 και θα ξεκινήσουν μόνο στους τομείς όπου μπορεί να καταδειχθεί ε, η αρχή της επικουρικότητας και μπορεί να ε, δομηθεί μέσα σε συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι θα πρέπει να ξεκινήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να κατατμηθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα είναι πάρα πολύ καλός αυτός ο, αυτή η περίοδος που μας δίνεται γιατί μπορούμε έτσι να ελέγξουμε πώς θα περάσουμε στις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, το δικό μου το προσωπικό στοίχημα είναι η συνοχή, ο δεύτερος πυλώνας της γεωργίας και η ε, έρευνα βεβαίως θα λειτουργήσουν, αλλά ε, ίσως να είμαι και λίγο απεσιόδοξη προς αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Νομίζω ότι είναι εφικτό αυτό που ζητούμε, κυρίως γιατί είναι μικρός ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, 1% του συνδυασμένου ΑΕΠ των κρατών μελών και δεν χρειάζεται να καλύψουμε μια, ένα ευρύ φάσμα δράσεων απέναντι σε όλες τις, όπως, μπορεί, όπως πρέπει να καλύψει ο εθνικός προϋπολογισμός. Το νέο αυτό ε, μοντέλο ε, μέχρι στιγμής δεν έχει ε, επιτύχει τίποτα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Δεν θα ήταν βέβαια η πρώτη φορά, η πρώτη φορά που το ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει το δρόμο για την δημόσια χρηματοδότηση. Να σας θυμίσω και τι γίνεται όταν τα κράτη-μέλη, όπου, σε περιπτώσει όπου τα κράτη-μέλη ακόμα μελετούν το κατά πόσο είναι εφικτό να ελέγξουν τους δικούς προϋπολογισμούς και τις ε, ε, μακροοικονομικές ε, παρατυπίες που υπάρχουν. Σας προειδοποιώ όμως, παρόλο που αυτό το σύστημα έχει τη δυνατότητα να σας δώσει τις λεπτομέρειες για την ποιότητα της δαπάνης, δεν θα είναι αυτόματο, εκτός και αν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη πρέπει να πάρουν την ευθύνη που τους ονολογεί και να παίξουν το ρόλο που πρέπει, να είναι διαφανή, ειλικρινή και να λογοδοτούν χωρίς απλούστευση των δημοσίων προμηθειών μιλήσαμε για τη Γενική Διάθεση ΜΑΡΤ, τα προγράμματα που λαμβάνουν κατά αποκοπή ποσά μπορεί να, πάρουν το, να ε, διατέχουν τον κίνδυνο να ξεπεράσουν τον προπολογισμό ή να μην επιτύχουν τους στόχους τους. Ε, Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Όταν μίλησα στην Επιτροπή ΣΟΥΡ για πριν από δύο χρόνια για το θέμα αυτό, με κατηγόρησαν ότι δεν ήμουνα ρεαλιστική και ότι ήμουν πολύ επαναστατική. Σήμερα ο κύριος Μουής ε, είπε ακριβώς ε, το ίδιο, ότι αυτή η προσέγγιση είναι επαναστατική. Άρα βλέπουμε ότι όντως η αλλαγή έχει αρχίσει ήδη να γίνεται. Thank you very much. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Και ίσως προς το τέλος της ημέρας αρχίζει να αναδύεται ένα επαναστατικό κλίμα. Ίσως μπορούμε πράγματι να αλλάξουμε το σύστημα και τώρα ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο για τα, από τα μέλη της Επιτροπής μας, ο κ. Μιλντερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί έπρεπε να απουσιάσω στο πρώτο τμήμα της ακρόασης. Υπήρχε μια άλλη κατεπίγουσα συνεδρίαση όπου θα έπρεπε να είμαι. Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία άκουσα και ιδίως αυτό που είπε ο κ. Μιλς και ότι η, κυρίως αυτό που είπε ότι το ελεκτικό συνέδριο είναι υποχρεωμένο να εκδώσει το πιστοποιητικό αξιοπιστίας με τον τρόπο που το κάνει μέχρι τώρα. Αναρωτιέμαι όμως αν για 18 χρόνια η καλύτε, τα καλύτερα μυαλά της Ευρώπης θεώρησαν ότι αυτή είναι η καλύτερη μεθοδολογία, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να το αλλάξουμε αυτό. Αν 27 από τα πιο εξέχοντα άτομα που προέρχονται από τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτή είναι η βέλτιστη μεθοδολογία, γιατί θα πρέπει να την διαφυσβητήσουμε. Βέβαια, πρέπει να την διαφυσβητήσουμε εάν πιστεύει κανείς ότι δεν είναι σωστή αυτή η μεθοδολογία και πιστεύω ότι υπάρχει γενική συμφωνία ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίνουν τη δική του αξιοπιστία, τη δική του δήλωση αξιοπιστία. Αυτό το έχει υποστηρίξει το Κοινοβούλιο. Το 2003 που ήμουν εγώ εισηγητή είχε τεθεί αυτή η διακρίκηση και την επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα φω στο τέλο του τούνελ. Πρέπει να είναι πολύ αμυδρό αυτό το φω, αλλά ενδεχομένω στου νέου δημοσιονομικού κανονισμού θα υπάρχει δυνατότητα εθελοντικά τα κράτη-μέλη να δίνουν μια εθνική δήλωση αξιοπιστίας. Το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να δούμε τώρα είναι γιατί τα κράτη-μέλη θα έχουν κίνητρο να κάνουν μια τέτοια δήλωση. Δεν πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόστιμα στα κράτη-μέλη εάν δεν το κάνουν αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πρόστιμα χωρίς να υπάρχει μια νομοθεσία την οποία τα κρατημέλη γενικά ούτε ή άλλως δεν θα δεχτούν. Πιστεύω δεν είναι ρεαλιστικό να βασιστούμε σε ένα εθελοντικό σύστημα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν κάποιο δόλωμα για τα κρατη που το κάνει <clears throat> ελκυστικό να υπάρχει αυτή η εθελοντική δήλωση, ίσως σε μειωμένη έλεγχη, ίσως το ωφέλιμα της αμφιβολίας για κάποια χρόνια. Αλλά αν έχετε κάποιες προτάσεις, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ιδιαίτερα καλόδεκτο γιατί η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο είναι πεπισμένοι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να κάνουμε πιο ελκυστικό για τα κάτι μελη να δέχονται αυτή την εθνική δήλωση αξιοπιστία. Οποιαδήποτε πρόταση είναι καλόδεκτη. Σα ευχαριστώ, Γιάν. Η κυρία Τσέσκοβα θέλει να λάβει το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω ερωτήματα, αλλά θέλω να πω ότι ο κύριος Σμουής το έθεσε το ερώτημα που είχα να θέσω εγώ και το απήντησε στην τόσο ενδιαφέρουσα παρέμβασή του. Και με, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την τόσο ενδιαφέρουσα παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα σχεδόν με όλα αυτά που ελέγξαν Ευχαριστώ. Και για πρωτού περάσουμε στο επόμενο σημείο θα ήθελα να ξέρω ποια είναι και η θέση της Κομισιόν για τα θέματα αυτά και ίσως το ερώτημα θα πρέπει να τεθεί προς τον κύριο Κράφτ και μετά θα δούμε πώς θα το επανασυνδέσουμε με τις ε, ε, αρχικές δηλώσεις όπως ανέφερε ο κύριος Γκρέι και ο κύριος Λέβη. Έχετε κύριε Κράφτ, κάτι να πείτε, είσαστε ικανοποιημένος με αυτά τα οποία έτεινε η κυρία Καλιολάιντ. Ναι κύριε Πρόεδρε, με ικανοποιούν ιδιαίτερα οι προτάσεις αυτές οι οποίες έχουν διατυπωθεί γιατί ανοίγουν τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη στοιχεία δημοσιονομικής διαχείρισης ως ένα συμπληρωματικό στοιχείο στο στοιχείο συμμόρφωσης μέσα στο πιστοποιητικό αξιοπιστία στον ΤΑΣ. Αν μου επιτρέπετε θα κάνω ένα περαιτέρω σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Μίλντερ γιατί και ο κύριος Μίλντερ αναφέρθηκε στα λόγια του κυρίου Μέης. Αν αρχίσω με το ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου, νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία ότι έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα συστατικά στοιχεία για την αποτελεσματική του λειτουργία. Δυστυχώς δεν λειτουργεί ακόμα αποτελεσματικά. Ελπίζω ότι η παρουσίασή μου ήταν σαφής για τα θέματα αυτά. Αν εφαρμόσουμε μηχανιστικά τυφλά τις πληροφορίες που μας δίνουν τα κράτη-μέλη, τότε το τελικό αποτέλεσμα θα είναι λαθασμένο. Γιατί τα κράτη-μέλη μας λένε τα ελέγχουμε όλα, όλα πάνε μια χαρά. Σε επίπεδο κομισιών και ελεκτικού συνεδρίου είναι, έχουν συμφωνήσει και τα δύο όργανα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το Κοινοβούλιο επίσης κατανοεί ότι είναι έτσι τα πράγματα και γι' αυτό επικρίνει, όπως φάνηκε και στην έκθεση απαραγής του κ. Γκάιερ Επομένως ε, θα πρέπει να ασκηθεί πίεση σε τεχνικό επίπεδο στα κράτη-μέλη και από το, Συμβούλιο, από το Ελεκτικό Συνέδριο και την Κομισιόν σε τεχνικό επίπεδο και από το Κοινοβούλιο σε πολιτικό επίπεδο για να υπάρχουν οι σωστές πληροφορίες. Γιατί νομίζω ότι μια σωστή διάγνωση κατάσταση είναι ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες δράσεις και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Από τη στιγμή που θα γίνει κάτι τέτοιο και που βγάζουν νόημα οι εθνικές δηλώσεις, λόγω πολιτικής πίεσης σε αυτούς οι οποίοι βραδιπορούν και δεν δίνουν τις κατάλληλες πληροφορίες. Αν δεν είναι αξιόπιστες αυτές οι πληροφορίες, τότε δημιουργούν όχι μόνο προβλήματα, αλλά και αντιφάσεις. Και κάποιο τότε θα πρέπει να είναι ο διαιτητής για να αποφασίσει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος από τους εμπειρογνώμονες μας θα ήθελε να λάβει το λόγο, ο κύριος Γκρέι. Να πω και εγώ κάτι σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν γίνει. Ναι, να αλλάξει συνθήκη. Η Κομισιόν το σκέφτηκε αυτό όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Αλλά δεν θα προχωρούσε αν δεν υπήρχε μια πρόταση του ελεκτικού συνεδρίου ή του Κοινοβουλίου αν υπάρξει αυτή η ανάγκη, το... αν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη το ελεκτικό συνέδριο να δίνει μια έκθεση για την κανονικότητα και την ε, ακρίβεια των λογαριασμών, τι θα μείνει πια από τις υποχρεώσεις του ελεκτικού συμβουλίου να ελέγχει τη, τα οικονομικά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πάει τότε το συνελεκτικό συνέδριο στην κατεύθυνση που ανέφερε η Επίσης, αν μιλήσουμε για απόδοση, ως πολιτική γνωρίζετε ότι αν έχουμε παραδείγματος χάρη μια γέφυρα στην ε, Σικελία που την φτιάνει η μαφία, εάν η Κομισιόν έλεγε δεν μας νοιάζει ποιος τη φτιάνει αλλά απλώς πρέπει να φτιαχτεί, θα είχαμε πολλά προβλήματα για την φήμη της Κομισιόν. Έχουμε δει λοιπόν στα διαφορετικά ταμεία πολλά προβλήματα όταν η Κομισιόν είχε χρηματοδοτήσει προγράμματα εμπορίας, προγράμματα σημών κατάρτισης, κατάρτισης και μας είπε το ελεκτικό συνέδριο δεν φτάνει να γίνουν τα προγράμματα κατάρτισης, πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καταρτίζονται και αν είναι ε, επιλέξιμοι για αυτά τα προγράμματα. Πρέπει λοιπόν να αναλάβει κανείς κάποιους κινδύνους ότι το πρόγραμμα μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση που ανέφερε η Κίστεν, αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να δούμε τους κινδύνους που ελοχεύουν. Δηλώσεις των κρατών μελών. Γιατί δεν το κάνουν, δεν κοστίζει τόσο πολύ. Μα σε ομοσπονδιακά κράτη όπως είναι η Γερμανία, η, η, Ισπανία, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σε κεντρικά κεντρική διοίκηση κράτη όπω είναι η Γαλλία, ίσω είναι πιο εύκολο. Αλλά σε ομοσπονδιακού χαρακτήρα ε, κράτη δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πάντα. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν εστιάζει ακόμα τις προσπάθειές της σε δηλώσεις από αυτούς που είναι πραγματικά υπεύθυνοι, είτε είναι οι φορείς που καταβάλουν τα χρήματα ή αυτοί οι οποίοι ε, ε τα ελέγχουν. Όλα αυτά πάντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και Θέλετε να λάβετε εσεί το λόγο. Μια-δυο κουβέντε, ίσω ο καθένα. Νομίζω η παρουσίαση του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν άκρο ενδιαφέρουσα. Απλώ να πω ότι αν δει κανεί την ιστορία του ελεγκτικού συνεδρίου και τι σχέσει του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δει το τι συνέβαινε με την νομοθεσία, Στην εποχή του ντελόρ. τα πράγματα ήταν τελείω διαφορετικά και αν κάνει μια σύνδεση με την διεθνή πραγματικότητα είναι διαφορετικά τα πράγματα στις Ηνωμένε Πολιτείες με τον κρατικό λογιστικό έλεγχο, με επιδόσεις περισσότερο παρά με συμμόρφωση ω κριτήριο. Με την πίεση ωστόσο υπήρχε το επικεντρικό σχόλιο ότι δεν υπήρχε αρκετός έλεγχος της συμμόρφωσης. Και εγώ ετοιμαζόμουν να πω κάτι παρόμοιο. Κάποιοι επικρίνουν τη θεωρία και την πράξη της δημόσιας διαχείρισης και της δημόσιας διοίκησης, διότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σαν κίνηση εκρεμούς που κάποια στιγμή να δίνει βάση σε κάποιες προτεραιότητες και όταν χρειάζεται σε κάποιες άλλες, δηλαδή τη συμμόρφωση και τις επιδόσεις ανάλογα με το τι είναι πιο σημαντικό η απομόνωση είναι φαίνεται η τάση που επικρατεί σήμερα, αλλά δεν είναι αυτός ο αποκλεισμός η απομόνωση η καλύτερη επιλογή. Δεν είναι απαραίτητο, όχι μόνο για τους λογιστές και τους εμπειρογνώμονε σε αυτό το τομέα, αλλά λόγω και κάποιων από τα στοιχεία της πραγματικότητας που συζητήθηκαν εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη όπως από, την, από τον κλάδο της λογιστικής μεν, αλλά τώρα έχουμε και μια ευκαιρία να μην επαφιόμαστε πλήρω σε τέτοιες εξειδικεύσεις. Οι λύσεις που χρειαζόμαστε δεν μπορούν να οριστούν μόνο από αυτή την κοινότητα. Πρόεδρος, ευχαριστώ και για να ολοκληρώσουμε ο κύριος Μουής πριν απαντήσετε κι εσείς, κύριε Καλιουλέιντ. Ναι, απλώς να τονίσω και να επικεντρωθώ στην ε, κρίση της Ευρωζώνης. Είναι σημαντικό για τους πολίτες μας να έχουν εμπιστοσύνη στα διάφορα της συστήματα που εφαρμόζονται. Είναι σημαντικό για τους πολίτες να μπορέσουν να κατανοήσουν το αρχιτεκτόνημα, την οικοδόμηση του συστήματος και ότι υπάρχουν ίσοι όροι παιχνιδιού για όλους. Αυτό και για τα εισοδήματα και για τα έσοδα και για τις δαπάνε, Εάν δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το μικροσκοπικό θέμα του μικρού ευρωπαϊκού υπολογισμού, πώς θα προχωρήσουμε και θα τονώσουμε την αμοιβή εμπιστοσύνη και όλα τα άλλα. Με την ε, κοινή οργάνωση των τραπεζικών μας συστημάτων, των δημοσιονομικών μας ε, συστημάτων. Αυτό είναι σαν να πηγαίνουμε μια βόλτα στην εξοχή σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη. Είναι ένα πικνίκ. Θα πρέπει κάπως εδώ να κατακτήσουμε τα κράτη-μέλη και να τα πείσουμε ότι πρέπει να αναλάβουν αυτά την υπογραφή του πιστοποιητικού αξιοπιστίας. Ε, πραγματικά εγώ καταντάω να αισθάνομαι ανόητος. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με μια στάση ενηλίκου στα κράτη-μέλη. Έχουν τους υπεύθυνους φορείς και θα πρέπει απλώς να κάνουν αυτό που κάθε φορολογούμενος απαιτεί. Είναι προϋπόθεση. Και ίσως να επιτρέψει να ανοίξει πόρτα για περισσότερη εμπιστοσύνη και εξοπιστία στο σύστημα συνολικότερα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μωής και πριν δώσω το λόγο στου, στην εισηγητρία και τι καταρκτικές τη παρατηρήσει, η κυρία Κάλιουλαϊντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κράτησα κάποια σημαντικά στοιχεία θεωρητικά και κάποιε παρατηρήσει των προηγούμενων ομιλητών και ήθελα να αντιδράσω. Δεν χρειάζεται να πάει κάνει στην ιστορία του ελεγκτικού συνεδρίου για να δει πώ έλαβε πολιτική σημασία. Ήταν αντίδραση σε μια από τι συστάσεις μέχρι τώρα για τις επιδόσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχει ένα πολύ ευαίσθητο όριο για το πώς πρέπει να δράσει ένα το ελεγκτικό συνέδριο ώστε να μην παρεμβαίνει στην όλη πολιτική διαδικασία. Δίνει γνωμοδοτήσεις για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού λόγου χάριου, αλλά παραμένει στα στενά όρια της άποψής του για τη συνοχή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Εάν ακολουθήσει κανείς την ε, κατεύθυνση της καταμέτρησης των επιδόσεων, θα πρέπει να μετατρόψει την συμμόρφωση σε επιδόσεις. Γι' αυτό και εγώ σήμερα έκανα αυτές τις ε, παρατηρήσεις. Διότι ίσω είναι πιο εύκολο να τα επιδιώξουμε αυτά από αυτά που έλεγε ο κύριος Γκρέι, δηλαδή αλλαγή στη συνθήκη. Επιδόσεις έναντι συμμόρφωσης δεν χρειάζεται να αλλάξει η συνθήκη για να αλλάξουν οι προϋποθέσεις των πληρωμών. Μόνο οι επόμενες περίοδοι προγραμματισμού. Οι δηλώσεις, δηλαδή τα πιστοποιητικά των κατομελών, είναι κάτι που αναφέρθηκε πολλές φορές στο ελεγκτικό συνέδριο της άποψης, ότι είναι καλό και χρήσιμο εργαλείο, αλλά το σημαντικό είναι ποιος έχει υπογράψει τις δηλώσεις και πώς γίνεται το, η δουλειά του ελέγχου για τις δηλώσεις αυτές. Αυτό αναφέρθηκε και για τις ε, εκθέσεις των νομοτήμων που κάποιος τις υπενήχθηκε εδώ πέρα, τις ετήσιες εκθέσεις. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να έχουμε αυτό το πλαίσιο, το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και χάρηκα που άκουσα και τις απόψεις των ακαδημαϊκών μας και των μεταπιστημιακών λένε ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορούσε να αλλάξει τον ορισμό του σφάλματος ή τη μεθοδολογία του. Ήταν μεταξύ των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν. Δεν είναι ότι δεν πίστηκε το ελεγκτικό συνέδριο να αλλάξει τη μεθοδολογία του και τον ορισμό, γιατί αυτό ήταν που μας είπε, υποχρέωσε να φτιάξουμε το σύστημα του ολοκληρωμένου εσωτερικού ελέγχου. Δεν είναι τέλειο ακόμη, δεν είναι τέλειο, αλλά ακολουθά τι αδρέ γραμμέ που σχεδιάσαν όλοι οι ομιλητέ που παρενέβησαν σήμερα στην ομιλία του. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ και τώρα λόγο στην συγκεκριά μα, την κυρία Τσέσκοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσω όλου του εμπειρογνώμονε, του εξπέρ, του προσκεκλημένου μα. Πραγματικά ήταν ε, πολύ πλούσιε οι παρεμβάσει σα, οι παρουσιάσει σα πολύ λεπτομερεί. Έχω να κάνω κάποιε παρατηρήσει για να κλείσουμε. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίστηκε πάνω σε συνθήκες συνθήκες μεταξύ των κρατών μελών ή συνθήκες μεταξύ διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό ακριβώς συζητούμε εδώ. Μιλούμε για ένα θέμα διαπραγμάτευσης, παρόλο που και αυτές οι διαπραγματεύσεις καμιά φορά τραβάνε σε μάκρος. Δεύτερον, πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε σωστά τα χρήματά τους. Αλλιώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο στο ελάχιστο θα έχει την ε, ε, δυνατότητα να διαχειρίζεται τα κονδύλια. Και τρίτον, υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά την οπτική τον, του πώς βλέπει κανείς τις, τους ισχύοντες κανόνες σε ό,τι αφορά την δήλωση αξιοπιστίας, τους κανόνες σε σχέση με το ποσοστό λάθους του 2%. Ερώτημα λοιπόν. Το πλαίσιο δαπανών θα πρέπει να το βελτιώσουμε, όπως προβλέπει ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός. Mm. Όλες αυτές οι πτυχές είναι διαφορετικές μεν, αλλά ε, συνδεόμενες και οι ε, διαφορετικές απόψεις που μας παρέθεσαν οι προσκεκλημένοι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και σε ό,τι αφορά το πλαίσιο ιστορικού ελέγχου. Ε, όλες αυτές τις παρατηρήσεις θα πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας για να δώσουμε και το σωστό μήνυμα από πλευράς Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τσέσκοβα, κυρία Συγήτρια. Εγώ μπορώ να υπογραμμίσω και να ε, αποδεχτώ πλήρως τα τελευταία σας σχόλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάρει τώρα την μπάλα. Αυτά τα οποία πρότεινε η κυρία Κάλιου θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι επαναστατικά αυτά που πρότεινε η κυρία Κάλιου αλλά υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο παραδείγματα που δείχνουν ότι είναι εφικτό αυτό. Εγώ ως βουλευτής σε περιφερειακό κοινοβούλιο στην Γερμανία είχα την ευκαιρία να δω ότι στον Καναδά, παραδείγματος χάρη, με μια αντικειμενική βάση προϋπολογισμού μπορεί να γίνει καλύτερος έλεγχος με μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορούμε φυσικά να τα μεταφέρουμε όλα αυτό, αυτούσια στην πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς θα εξασφαλίσουμε την πολιτική θέληση για μια τέτοια αλλαγή. Όλα αυτά τα στοιχεία και οι συμβολές των ε, εμπειρογνωμόνων. Μας έχουν δώσει πολλές ιδέες και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και τις ομιλήτριες. Ίσως ήμουν λιγάκι αυστηρός και αναγκάστηκα να είμαι αυστηρός για την διαχείριση του χρόνου, αλλά νομίζω ότι μέσα στο χρόνο που είχαμε μπορέσαμε με τη βοήθειά σας να διεκπαιρεώσουμε όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ και κλείνει λοιπόν η συνεδρίασή μας. Διακόπτουμε μέχρι αύριο και καλό τους συντονιστές να παραμείνουν για την συνάντηση των, των συντονιστών απόψε. Ευχαριστώ και τις μεταφράστες που μας έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα και τη γραμματεία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και του Ελεκτικού Συνέδριου. Ευχαριστώ.